Ο, ο Πρόεδρος. Καλώς ορίσατε. Σας ε, ευχαριστώ που ήρθατε. Και κυρίως να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τον κύριο Σαβίσκια, ο οποίος προγραμμάτισε όλες αυτές τις συναντήσεις για την μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και θα προχωρήσουμε σε αυτές τις επαφές την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Έχουμε τη σημερινή ευρωπαϊκή εκδήλωση, ε, την οργανώσαμε εμείς και έχουμε τώρα τους ε, εισηγητέ οι οποίοι θα μας ε, δώσουν τα φώτα του απόψε. Οπότε πρόκειται να προχωρήσουμε επομένω σε μια τέτοια επικοδομητική συζήτηση και για, τις, για τους τρεις για τρία θεσμικά όργανα τα οποία αφορούν την ρύθμιση τη ΚΑΠ και έτσι θα αποδείξουν, τα στείλουμε ένα μήνυμα το οποίο θα αφορά την πρόθεση συνεργασία. Ελπίζω ότι τελικά θα έχουμε ε, μια ποιότητα στη σημερινή ε, συνάντηση που θα είναι στο ύψο των προσδοκιών των Ευρωπαίων και βεβαίω ελπίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση, θα δοθούν απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα τα οποία εκκρεμούν και που έχουν ε, σχέση με προβλήματα τα οποία έχουν ξεκινήσει από το παρελθόν και εδώ το κοινοβούλιο μας θέλει να εξετάσει τι γίνεται με αυτήν τόσο σημαντική μεταρρύθμιση. Αυτή η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει μέσα σε αυτήν την ε, εξαιρετικών συνθήκων συγκυρία. Και αυτό διότι υπάρχει ορίζοντας δεδομένος, υποχρεωτικός, δεσμευτικός. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ότι πολλοί λένε ότι ξεκινά μια νέα εποχή για την ε, γεωργία και όσον αφορά τα θέματα τα αναπτυξιακά και εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την διατροφική επάρκεια και επομένως πρόκειται για ε, να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τους πόρους όσον αφορά τι γίνεται μεταξύ βορρά και νότου και επίσης αυτός ο αγροδιοτροφικός τομέας ε, έχει γνωρίσει μεγάλες αλλαγές και οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τη συνέχιση των επιχειρησιακών, των επιχειρηματικών, των οικονομικών πτυχών του θέματος, τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επίσης να δούμε και πώς θα συνεχίσει υπάρχει συνέχεια και συνέχιση όσον αφορά τη μεταποίηση. Θα πρέπει επίσης να μπορεί ο κλάδος να παράσχει τις σχετικές εγγύσεις στους Ευρωπαίους καθαλωτές, ούτως ώστε εκείνοι να μπορούν να έχουν κάποιες εγγύσεις ποιοτικέ ε, για κάποια είδη διατροφής τα οποία να είναι υγιεινά. Και αυτό αφορά το κοινωνικό μας τελικά μοντέλο, το ευρωπαϊκό. Επομένω αυτό αφορά και τους εργαζόμενους, ε, αφορά τους Ευρωπαίους, αφορά το τι θα γίνει με τα δημόσια αγαθά, τι θα γίνει με την κοινωνική συνοχή. Εδώ και πολλά χρόνια τα λέμε αυτά. Και πρόκειται για μία από τις πιο βασικές φιλοδοξίες της Ευρώπης στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε σε σχέση με κάποια βιώσιμη γεωργία, αηφόρο και να δούμε με ποια μέσα πολιτική θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την πρόκληση του σήμερα. Πώς θα μολύνουμε λιγότερο το περιβάλλον αλλά θα μπορέσουμε να παραγαγούμε περισσότερο και ωστόσο να δούμε το ότι υπάρχουν εδώ, ελοχεύουν εδώ πάρα πολύ σημαντικοί κίνδυνοι. Για μας αυτό είναι βασικό θέμα ουσίας. Αυτό θα είναι ο μπούσουλας για το πώς θα προχωρήσουμε. Επομένως, με πνεύμα συνεργασία τα θεσμικά όργανα τώρα θα προχωρήσουν σε αυτή τη μεταρρύθμιση και ελπίζουμε ότι θα ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσει αυτού του νέου στόχου. Επίσης θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε συμμόρφωση προς την συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή ότι η κοινή αγροτική πολιτική αφορά τη διαδικασία της συναπόφασης. Θα πρέπει επομένω να ληφθεί υπόψη ότι έτσι θα εκπροσωπηθούν πιο άμεσα οι πολίτες για τη λήψη των αποφάσεων. Σε αυτή τη διαδικασία επομένω θα πρέπει να δούμε μια καινούργια αξία, θα πρέπει εδώ να εκτιμήσουμε την ε, συμβολή της ε, Προεδρίας. Προχώρησε και αυτή η δέσμη των μέτρων για τα γαλακτοκομικά. Αυτό έγινε σε πρώτη ανάγνωση και έτσι με αυτή την διαδικασία της συναπόφασης θα βελτιώσουμε τις προσθήκες της, ε, συγγνώμη, της, τα, τα όσα θέλει τώρα να εισφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επομένως τα κείμενα αυτά τα οποία μας δίνουν ένα χάρτη πορεία στον οποίο θα μείνουμε πιστοί. Πρόκειται για το έργο του που θα επιτελέσουμε στους επόμενου επόμενους μήνες και όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Κατά αυτό το έργο του που θα επιτελέσουμε και επομένως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η ΚΑΠ, η μελλοντική, να είναι πιο ευέλικτη, πιο αποτελεσματική, να μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις που δυστυχώς τώρα μαστίζουν τις αγορές και τον κλάδο βεβαίω αυτών. Οπότε παρακαλούμε ο κύριος Επίτροπος να μας βοηθήσει στο έργο μας και έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία των νωρίτερο δυνατόν. Με αυτή τη συμφωνία θα πετύχουμε, ελπίζουμε, τους κοινού στόχους. Θα απλουστεύσουμε τα μέσα ευελιξίας και θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν με κάποια μέτρα πολιτικής, ε, με πολιτικές ε, που σηκώνουν πολλή συζήτηση. Θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Αλλά το επιθυμητό είναι να πετύχουμε αυτό το στόχο και έχουμε επομένως μία νέα γενιά γεωργών οι οποίοι έχουν κάποιες προσδοκίες και επομένως θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία όχι μόνο με τα θεσμικά όργανα, με τις αρχές αλλά θα πρέπει οι γεωργοί να συνεργαστούν και με την υπόλοιπη κοινωνία. Όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Σήμερα θα δουλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα και ελπίζουμε οι συγητές να μας βοηθήσουν όπως πρέπει. Πάντως, μέχρι ότου καταλήξουμε στο τι θα γίνει με τις δημοσιονομικές προοπτικές, Νομίζω ότι το να κατεβάσουμε τροπολογίες και να κάνουμε ψηφοφορίες δεν ωφελεί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η αρχιτεκτονική του οικοδόμου μήματος που να κάνουμε, πώς θα έχει αυτό στέρεα θεμέλια. Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει και κάποια τεχνικά, τεχνοκρατικά σημεία. Νομίζουμε ότι αυτή η οικολογική άποψη, το δεύτερο πυλώνα, η έννοια του ενεργού γου ενεργητικού γεωργού, όλα αυτά είναι θετικά. Όλα αυτά τα έχουμε αναφέρει, συζητήσει, θα εμβαθύνουμε, θα πρέπει να ζητήσουμε νέους δρόμους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και με την τόσο αξιόλογη συμβολή των ε, προσκεκλημένων μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Επιστημονική Κοινότητα, πιστεύουμε ότι η εκδήλωσή μας θα πετύχει. Εγώ είμαι πανεπιστημιακός που τώρα έχω μπει στην πολιτική και γι' αυτό σας λέω ότι έχω την πεποίθηση ότι ακριβώς όπως έγινε και στο παρελθόν θα μπορέσουμε επικοδομητικά να εργαστούμε κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό και για τους Ευρωπαίους αλλά και για τους Γεωργούς εφόσον όλους και τώρα δίνουμε τις κοιτάλες στον κύριο σε τον τον ε, Επίτροπο. Ευχαριστώ Πάολο. Ευχαριστώ, Παύλο. Σήμερα χαίρομαι διότι συμμετέχω στην τρίτη συνάντηση στα πλαίσια των ε, τριών συνεδριάσεων που είχαμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε από κοινού με την ε, Πολωνική Προεδρία. Από κοινού, τα τρία θεσμικά όργανα, μετά από την νομοθετική πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργάνωσε σε αυτή την ίδια την αίθουσα μία διάσκεψη όπου έγινε συζήτηση με τους Υπουργούς Γεωργίας και την Κομισιό. Η Πολωνική Προεδρία πρόσφατα επίσης οργάνωσε και μια άλλη διάσκεψη με τις διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα της Γεωργίας καθώς και με το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών και η Επιτροπή όπως είχε υποσχεθεί σήμερα προτείνει να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από τις αναλύσεις που έγιναν και τις παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν οι εμπειρογνώμονες και οι δήμονες στα πλαίσια αυτής της νέας μεταρρύθμισης. Με αυτή λοιπόν τη διάσκεψη σήμερα σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση που είναι η βάση της εμβάθυνσης αυτών των προτάσεων. Σα είπα ευθύ εξ αρχή ότι είναι συνεκτικέ όλε αυτέ οι προτάσει, δεδομένου ότι αφορούν το σύνολο τη κοινή αγροτική πολιτική Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μετά από την πρώτη παρουσίαση. Εγώ είπα ότι χρειαζόμαστε χρόνο για να εμβαθύνουμε πραγματικά στις προτάσεις και να κάνουμε τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων ιδεών που συμπεριλαμβάνονται στην πρόταση αυτή για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στις συμπεράσματα και να κάνουμε και αναλύσεις και κριτικές και επικρίσεις ίσως. Κάποιους μήνες λοιπόν μετά από την κατάθεση της πρότασης πρέπει να πω ότι όπως είπε και ο Πάολο είχαμε συζητήσει ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται εμβάθυνση των προτάσεων αυτό και του περιεχομένου τους έγιναν στις ε, ομάδες εργασίας που οργανώθηκαν σε επίπεδο Συμβουλίου επίσης και κάποιες ε, ενδελεχείς συζητήσεις και τώρα μπορούμε με διαφορετική ματιά αν θέλετε και με πιο συγκεκριμένο τρόπο και με μεγαλύτερη ακρίβεια να δούμε περί τίνος πρόκειται. Ο επιστημονικός κόσμος και οι εμπειρογνώμονες, όπως ξέρετε, συμμετείχαν σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία προτάσεων για τη μεταρρυθμίση ευθύ εξ αρχής. Δεδομένου ότι στην προπαρασκευαστική φάση και στην δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε πέρυσι, βασιστήκαμε πάρα πολύ στις ιδέες που κυκλοφόρησαν δημοσίως και ανελήφθησαν από τις, ε, από τις διάφορες ομάδες εμπειρογνωμόνων, ειδημόνων και οικονομολόγων και η επιστημονική κοινότητα συμμετείχε σε όλες τις αναλύσεις τις οποίες οργάνωσαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής για τις μελέτες επιπτώσεων αυτής της μεταρρύθμισης για να μπορέσουμε πέραν των πολιτικών αποφάσεων να βασίσουμε τις προτάσεις μας σε αναλύσεις συγκεκριμένες και σε συμπράσματα στα οποία κατέληξαν οι μελέτες σκοπιμότητας και επιπτώσεων. Σήμερα τι κάνουμε. Δίνουμε μία άλλη προοπτική στις διάφορες προτάσεις βασιζόμενες στις αναλύσεις που έγιναν και έτσι θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο των διαφορών προτάσεων, αλλά θα τις δούμε και σε μια άλλη προοπτική, σε μια ευρύτερη προοπτική από αυτήν που αφορά αμυγός τους μηχανισμούς της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δεν θα πρέπει παρόλα αυτά να εξηγούμε, πέραν όλων αυτών των αντικειμενικών αναλύσεων, τι οποίε χρειαζόμαστε πάντα όταν είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αποφάσει, ότι πολλέ φορέ μεταξύ του επιθυμητού και του εφικτού υπάρχουν διαφορές. Και υπάρχει και μια πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρόκειται λοιπόν για στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και πάντα θα πρέπει να καταλήγουμε σε, μια σε ένα συμβιβασμό βάση αποφάσεων, δηλαδή να ακολουθούμε πάντα την μέση οδό, τη χρυσή τομή από ε, πολιτική σκοπιά και από τι προβάσει των διαθέσιμων κονδυλίων στον προπολογισμό. Στα πλαίσια αυτή τη νομοθετική πρόταση υπάρχει ένα στοιχείο κλειδί, το οποίο φαίνεται και από όλε τι επιστημονικέ αναλύσει. και είναι η ανταγωνιστικότητα τη κοινή αγροτική πολιτική. Σε αυτά τα πλαίσια όχι μόνο πρέπει να παράγουμε περισσότερο, αλλά καλύτερα και βασιζόμενοι στους μία περιόριστους πόρους που διαθέτουμε. η εσωτερικοποίηση των αναγκών μας όταν μιλάμε για καλή διαχείριση των πόρων είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας. Διότι η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι αηφόρος και ο μηχανικισμός που θα θέσουμε σε εκείνη για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή την αηφορία θα πρέπει να γίνει κατανοητός και να γίνει αποδεκτός από αυτούς που παρέχουν τους πόρους, δηλαδή το χρήμα. Προσπαθήσαμε λοιπόν βάσει όλων αυτών των στοιχείων να κάνουμε μία σωστή πρόταση. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε νέες προοπτικές στους γεωργούς και στους παραγωγούς σε σχέση με τις αγορές, σε σχέση με την ε, γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται. Διότι όλο και περισσότερο η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας θα πρέπει να γίνεται κυρίως σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία σήμερα έχει διευρυνθεί όλο και περισσότερο με, όλο και περισσότερο με κράτη μέλη στα οποία θα πρέπει οι αγρότες να γίνουν οι πρωταγωνιστές του επαγγελματικού, του οικονομικού και κοινωνικού τους μέλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι γίνει να γίνει με τη συνδρομή των επαγγελματικών οργανώσεων των γεωργών και αυτό το αναφέρουμε, είναι σημαντικό στοιχείο για να ενισχύσουμε τη ε, ε, σημασία τους αλλά και βασιζόμενοι ο καθένας στο γεωγραφικό περιβάλλον στο οποίο είναι κανένας. Δεδομένου ότι ό,τι γίνεται σε επίπεδο γεωργίας έχει σχέση με το μέρος στο οποίο βρίσκεται ο γεωργός και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό τον ε, δεσμό με τον ύπεθρο, ε, τον χώρο στον οποίο αναπτύσσει η δραστήριο του ο Γεωργός, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις άλλες κοινοτικές πολιτικές που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και να συντονίσουμε τις πολιτικές μας. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία ήθελα να σας υπενθυμίσω. Μετά την παρουσίαση που θα γίνει από τον ε, υπεύθυνο της Πολωνικής Προεδρίας, θα κάνει τον συντονισμό της συζήτησης ο κύριος Σίλβα Ροντρίγκε, Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Θα ακούσουμε τους συμπεριγνώμενες και μετά θα κάνουμε την συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, την Πολωνική Προεδρία και κυρίως τη Δανέζικη, η οποία ακολουθεί, δεδομένου ότι εκείνη θα κληρονομήσει όλη αυτή την διαδικασία. Και κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Βεβαίως, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχει στενά σε όλη αυτή τη δικασία και με την αγαστή συνεργασία μεταξύ μας πιστεύω ότι θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και έγκαιρα ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη και οι αγρότες να χρησιμοποιήσουν το συντομότερο δυνατό τη νέα αυτή κοινή αγροτική πολιτική έτσι όπως θα την ε, μεταρρυθμίσουμε. Δίνω τώρα το λόγο αμέσω στον κύριο Μάρεκ Σαβίνσκι, πρόεδρο του Προεδρεύοντο Συμβουλίου σε θέματα γεωργίας και αλίας, Υπουργό Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου της Πολωνίας. Σας ευχαριστώ. Panie i panowie profesorowie, drodzy Κυρίες και κύριοι, κύριοι καθηγητές, πυρογνώμονες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο Ντεκάστρο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι, διότι τελικά ανέλαβαν την πρόκληση του να γίνει αυτή η συζήτηση για την μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Σα υπενθυμίζω ότι στι 7 Νοεμβρίου ξεκίνησε αυτό ο κύκλο των επαφών μεταξύ μα. Ξεκινήσαμε με την αγόρευση του Πρόεδρου Μπούζεκ. Κατόπιν συνεχίστηκε και ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων όλων. Και τώρα έχουμε και τους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, οπότε και εγώ δεν μπορώ παρά να τονίσω ότι από όλο το επιστημονικό στερέωμα έχουμε τώρα εκπροσώπους. Και έτσι, με δυναμικό τρόπο, συνεχίζεται η προσπάθεια του Ντάτσιαν Τσόλος του κυρίου Επιτρόμπου. Επίσης, έχουμε συγκροτήσει και νομοθετικές ομάδες που εργάζονται συνεχώς. Βεβαίως και είναι κάτι απαραίτητη αυτή η διαδικασία, διότι μέσα από αυτή τη διαδρομή νομίζω ότι όλοι θέλουμε να υπάρξει μια εις βάθος αλλαγή θα πρέπει μακρόπνο να δούμε τις διαστάσεις της γεωργικής μας πολιτικής. Να δούμε τι θα γίνει με τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Τι θα γίνει με την στρατηγική 2020. Θα πρέπει να δούμε ακόμη πιο δύσκολο τι θα γίνει για τον ορίζοντα του 2050. Είμαστε υποχρεωμένοι επομένω να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις για τις υπάρχουσες ανάγκες. Είμαι θα πεπισμένη ότι με την μεταρρύθμιση αυτή η οποία μόλις τώρα ξεκίνησε θα καλύψει αυτά τα οποία θέλουμε. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή αυτής της διαδρομής οπότε και η επιστήμη, η ευρωπαϊκή επιστήμη θα μας δώσει απαντήσεις. Θέλουμε τώρα να δώσουμε κάποιε απαντήσεις, δηλαδή το τι θα γίνει με κάποιο είδους τέτοιες μακρόπνες προοπτικές, πώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και να μπορέσουμε να καλύψουμε τις σχετικές ανάγκες οπότε και γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον να δούμε με ποιους τρόπους θα καλυφθεί ο προϋπολογισμός για τον οποίο βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όμως θα πρέπει να δούμε ότι η Ευρώπη σήμερα δεν έχει τόσα περιθωρία ελιγμών υπό την σημερινή συγκυρία. Άρα, σήμερα έχουμε αυτές τις τρεις θεματικές ενότητες που θέλουμε να συζητήσουμε και επομένως έτσι θα αναδυθούν κάποια ερωτήματα να δοθούν κάποιες ε, απαντήσεις και να αναζητηθούν κάποιες λύσεις. Διατροφική επιστηστική ασφάλεια, να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα θέματα ανταγωνισμού, αυτά τα οποία μας απασχολούν εδώ και πολύ καιρό. Το 2008 έγινε μια πρώτη προσπάθεια μεταρρύθμισης και θεωρήθηκαν ότι αυτά τα ζητήματα είναι θέματα προτεραιότητας. Επίσης, ε, αυτό που μας προσφέρει δεν είναι μόνο τα ποσοτικά θέματα, αλλά μετά στην πρώτη προσπάθεια μεταρρύθμισης που έγινε το 2003 έγινε αντιληπτό ότι η πιστιστική ασφάλεια είναι επίσης σημαντική όσον αφορά και την ποιοτική της πτυχή. Γιατί θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να φροντίσουμε, να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Και γι' αυτό και οι γεωργοί μας έχουν ευξημένα και πιεστικά καθήκοντα όσον αφορά αυτό το στόχο, το περιβάλλον. Θα πρέπει επομένω να φροντίσουν τα παράπλευρα ούτως θέματα αλλά χωρίς και να παραμελούν το κύριο θέμα, το κύριο καθήκον που είναι η παραγωγή. Βεβαίως βροχή είναι τα παράπονα του Ευρωπαίου όσον αφορά την τιμή των αγροτικών προϊόντων. Αλλά ταυτόχρονα και οι γεωργοί παραπονούνται ότι το εισόδημά τους σε σχέση με το τι κόπο καταβάλουν είναι μικρό. Έχουμε εμείς από πλευράς μας κάποιες επιτροπές σε ψηλό επίπεδο που προσπαθούν να καλύψουν τα προβλήματα της ε, διατροφικής αλυσίδας όμως αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερο πολιτικό θάρρος, περισσότερη βούληση, ούτως ώστε αποφασιστικά να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Γιατί και η επιστήμη αλλά και η οικονομία έχουν πολλές προτάσεις. Πολλές προτάσεις που δίνουν απαντήσεις, προτείνουν ενδείξεις που μας βοηθούν σε σχέση με το τι επιλογές θα κάνουμε για λύσουμε των προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Άρα χρειάζεται μια ισόρροπη, διαρκής, σταθερή ανάπτυξη. Να δοθεί μια νέα σύλληψη στην γεωργική πολιτική. Πώς θα έχουμε καθαρό περιβάλλον να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Διαρκώς αλλάζουμε τα πλητές που περιβάλλον αλλά και την παραγωγή. Έχουμε την Επιτροπή για την Πράσινη Πολιτική και θα πρέπει να δούμε το πώς θα κάτσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό του τι πετύχαμε μέχρι σήμερα και να δούμε και τι χρειάζεται να κάνουμε. Πώς θα προτείνουμε κάποιες λύσεις για τις ε, ζωοτροφές, για την ισορροπημένη γεωργία και επίσης πώς θα δοθεί συνέχεια στις οδηγίες που αφορούν το περιβάλλον. Προχωρούμε σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης προς τις ίδιες κατευθύνσεις αλλά πρέπει να σκεφτούμε και το ότι τους έχουμε δώσει βαριές ευθύνες τώρα των Γεωργών και άρα θα πρέπει να αναλύσουμε το πώς θα προχωρήσουμε σε αρμονία με το περιβάλλον και πώς θα δοθούν κάποια οικονομικά κίνητρα στη Γεωργία. Τι θα γίνει με τους ε, όλο ένα και περισσότερες απαιτήσει που τάσσονται στην γεωργική παραγωγή. Να μην ξεχνούμε ότι οι χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετική αφετηρία και διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετική προϊστορία και αν θέλουμε σήμερα να έχουμε ομοιογενή, ισορροπημένη ανάπτυξη παντού στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα. Η γεωργική πολιτική με τις δεδομένες ε, ε, επιδοτήσεις αξιοποιεί τις δυνατότητες που υπάρχουν τα μέσα τα οποία έχει η γεωργική πολιτική ιστορικά σε σχέση με την ιστορική της παραγωγή, σε σχέση με την παραγωγή τροφίμων. Μπορεί η γεωργική πολιτική να συνεχίσει να παρέχει τις εγγυήσεις που ζητούμε και ταυτόχρονα να σέβεται το περιβάλλον πάντοτε χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να πετύχουμε κάποιες αξιόλογες επιδόσεις. Μπορούμε με τον προβληματισμό το οποίο έχουμε αναπτύξει να αποστασιοποιηθούμε από αυτή την παράδοση της οικονομικής στήριξης που σέρνουμε πίσω μας. με τη δεδομένη δημοσιονομική προοικοδότηση πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις και την παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Δεν θέλω τώρα να κατηγορήσω τους προκατόχους μου, αλλά συζητούμε τώρα για τον προϋπολογισμό της Γεωργίας, για τη μεταρρύθμισή της, που αλλά δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε αυτήν την ε, μεταρρύθμιση μέσα στα στενά ενό συγκεκριμένου προϋπολογισμού. θα πρέπει να δούμε πέρα από τον προπολογισμό αυτόν για να δούμε πώς θα καλύψουμε τις προσδοκίες γεωργών και καταναλωτών. Επίση θα πρέπει να δούμε ότι και αυτή η χρηματοδότηση έχει κάποιο όριο στον αφορά το τι χρηματοδοτεί, τι στηρίζει. Μήπως θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο ανταγωνισμό, μήπως θα προσέξουμε περισσότερο ανάπτυξη. Νομίζω ότι η επιθυμητή ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω των ενεργών, δυναμικών, ενεργητικών γεωργών. Και έτσι θα πρέπει να γίνει η κατανομή των, πόρων των μέσων πολιτικής έχουμε. Με αποφασιστικό τρόπο, ότι μέσα στα πλαίσια τη κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να ενισχύσουμε τον δεύτερο πυλώνα σε σχέση με, με τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη. Εάν δε πραγματικά θέλουμε να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη η Ευρώπη, τότε πρέπει να δούμε πώς θα καλύψει τις ευαισθητικές ανάγκες και οπότε αν το θέλει αυτό η Ευρώπη θα πρέπει, λέω, να μεταρρυθμίσει, να αναθεωρήσει την γεωργική της πολιτική. Εν κατακλείδη κυρίε και κύριοι, αυτό το οποίο θέλω είναι να μας δώσει η επιστήμη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Δηλαδή το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον υπάρχοντα προπολογισμό, τις υπάρχουσες δημοσιονομικές δυνατότητες και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια γεωργική πολιτική η οποία να καλύπτει όχι μόνο την παραγωγή αλλά και ανάπτυξη και ανταγωνισμό. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε στις επιδόσεις μας σε σχέση και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ. Ε, Μάρεξ, ευχαριστούμε λίγο πρόεδρο. Και τώρα. Έχω δίνω το λόγο στον Γενικό Διευθυντή της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης για την Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπέθρου ή στον <clears throat> κύριο Σίλβα Ροντρίγκε. Και μετά θα έχουμε ελπίζουμε αρκετό χρόνο ώστε να γίνει συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κάστρο, ευχαριστώ τον κύριο Τσόλο και κύριε Σαβίσκη που μου δίνετε τη δυνατότητα να συντονίσω την συζήτηση του απογεύματος. Έχουμε τρεις διαφορετικές ενότητες να εξετάσουμε μαζί για να ακούσουμε τους ε, εμπειρογνώμονες για κάθε ένα από τα θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Κάθε ε, εμπειρογνώμων θα μιλήσει για 10 λεπτά και μετά θα έχουμε για μισή ώρα στο τέλος των ε, παρεμβάσεων συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, θα ζητήσω στον κύριο Τζοβάνι Ανανία ε, του Πανεπιστημίου της Καλαβές στην Ιταλία και τον κύριο, από τον κύριο Ερβέγγι Γιωμάρ του Εθνικού ε, Ιδρύματος Έρευνας της ε, Γεωργίας από τη Γαλλία να μας μιλήσουν για την ασφάλεια των τροφίμων την και την ανταγωνιστικότητα της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Επαναλαμβάνω 10 λεπτά ομιλία ο καθένας και μετά μισή ώρα συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντικό και μια μεγάλη πρόκληση. Πάνω από 15% του παγκοσμίου πληθυσμού ε, υποσυτίζονται σήμερα. Όμως, αφήνοντας κατά μέρο τις επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης, της επιστημιστικής, έχει αλματοδός αυξηθεί ο πληθυσμός παγκοσμίως. Και έτσι ακριβώς έχουν αυξηθεί και τα αριθμητικά στοιχεία και των κατοίκων του αναπτυσσόμενου κόσμου και του αριθμού των υποσυτιζόμενων μεταξύ του 1970 και σήμερα. Αριστερά βλέπετε τους υποσυτιζόμενους και δεξιά βλέπετε το ίδιο στοιχείο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η επιστημιστική ασφάλεια ε, έχει, διακυβεύεται αυτή τη στιγμή λόγω ακριβώς της δημογραφικής έξαρσης και αύξησης 34% ε, ενώ ε, η θερμιδική ε, παροχή ανακάτοικο χρειάζεται να αυξηθεί κατά 26,2%. 2.000 ε, θερμίδες χρειάζονται για μία υγιή διατροφή, αλλά το 26% ε, του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε αυτή τη διατροφή. Γι' αυτό λοιπόν όταν ε, κάνουμε μία περιφερειακή αξιολόγηση των επισητιστικών αναγκών αντιμετωπίζουμε αυτές τις τεράστιες προκλήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Εφόσον λοιπόν η, ε, παρόλο που έχει αυξηθεί ο πληθυσμός αλματοδό στην Ιφίλιο, η επάρκεια των τροφίμων θα μπορούσε να λειτουργεί ικανοποιητικά εάν υπήρχε ίσως καταμερισμός του πληθυσμού στις διάφορες υπήρους και με ίση οικονομική ανάπτυξη. Όμως δυστυχώς ένας από τους 7 ε, κατοίκους της υφηλίου ε, μας υποσυτίζεται. Και το πρόβλημα, δηλαδή 925 εκατομμύρια υποσυτίζονται μονίμως. Το πρόβλημα δεν είναι η ανεπάρκεια της ε, προμήθειας τροφίμων, αλλά τα προσκόμματα στην πρόσβαση στα τρόφιμα, κυρίως η φτώχεια. Σήμερα το πρόβλημα το μεγάλο είναι η φτώχεια, όχι η έλλειψη τροφίμων. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε σαφή ευθύνη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας. Η επισητιστική ασφάλεια στην Ευρώπη είναι ένα πρόβλημα, το οποίο έχει άμεση επίπτωση βεβαίως στις φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού. Και αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από την πολιτική της ΚΑΠ, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια διατομεακή πολιτική, η οποία θα εγγυηθεί η ισότιμη πρόσβαση στις ε, πηγές ε, και στα προϊόντα, τα επισητιστικά τα οποία χρειάζονται είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο να διευκολύνουμε την πρόσβαση στα, τρόφιμα. Εάν δούμε τι προοπτικές διαγράφονται για την επιστημιστική ασφάλεια, υπάρχει μια τεράστια πρόκληση και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα σταθερό βαθμό ανάπτυξης επισητιστικής επάρκειας και προμηθειών έτσι ώστε να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με σταθερά ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης. Η παραγωγή τροφίμων τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν μας επιτρέπει αισιοδοξία. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ο μέσος όρος της ετήσιας ε, προσόδου Τη ετήσια απόδοση σε καλαμπόκι, ρύζι και δημητριακά. 63 με 2005. Βλέπετε λοιπόν σταθερή μείωση ε, των αποδόσεων για τα τρία αυτά βασικότατα προϊόντα. Γιατί? Διότι έχει μειωθεί το ποσοστό επενδύσεων, ε, μια φθήνουσα, σταθερά φθήνουσα πορεία, και αυτή η φθήνουσα των αποδείσεων έχει προφανώς οδηγήσει στην μείωση ε, του μέσου όρου ετήσιας απόδοσης ε, των τριών αυτών ε, βασικών προϊόντων. Τώρα, τι επενδύσεις χρειάζονται, τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί η φτώχεια και να διασφαλιστεί η επισητιστική επάρκεια, η επισητιστική ασφάλεια. Σας είπα, μείωση της φτώχειας. Αυτό είναι το υπαρθμόν ένα στοιχείο που πρέπει να πολεμήσουμε ε, με κάθε μέσο. Βέβαια, αυτό δεν είναι το μόνο μέτρο, το μόνο πρόβλημα που μας απασχολεί. Μπορούμε να κάνουμε και διάφορα άλλα ε, πράγματα μέσω βελτιωτικών πολιτικών. Καταρχάς πρέπει να εδραιώσουμε πολιτικές στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι οποίες ενισχύουν την ε, αγροτική παραγωγή και δεν τη βλάπτουν. Δεν είναι δηλαδή ε, ζημιογόνες. Δεύτερον, πρέπει να διευρύνουμε τις επενδύσεις, οπωσδήποτε, και δει τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό είναι κυρίως μια ευθύνη της διεθνούς κοινωνίας ε, για την στήριξη της αηφόρους ανάπτυξη ε, της παραγωγικότητας, για την μείωση των, του κόστους παραγωγής, για την βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και για την υποστήριξη των ε, καινοτοπιών. Εξετάζοντας τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, με αναλυτικό φακό, δεν μπορούμε άμεσα να διαπιστώσουμε όλες αυτές τις ανάγκες ε, ανατομέα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ε, και με τη βοήθεια της ε, ανακοίνωσης της Κομισιόν για το νέο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής εντοπίσει τα βασικά στοιχεία, τις βασικές πτυχές ε, προς τις οποίες πρέπει να προσανατολιστούμε. Υπάρχουν Καταρχάς, ε, με ε, σαφής ανάγκη να ενισχύσουμε την ΚΑΠ και τον μηχανισμό μεταρρύθμισης. Αλλά για, κατά τη δική μου ε, άποψη, αυτά τα επιχειρήματα δεν αναφέρονται μόνο στην ΚΑΠ και στη μεταρρύθμισή της. Πρέπει να αναπροσανατολίσουμε την αγορά. Επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε την ΚΑΠ, δεδομένου ότι έχει υποβαθμιστεί και έχει φθαρεί για την πάροδο των ετών. Αυτό Δηλαδή, ε, ο αναπροσανατολισμός των αγορών και η στήριξη των φθηνουσών στοιχείων της ΚΑΠ σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και τα στρατηγικά μέτρα. Επίσης, 30% του προϋπολογισμού της ΚΑΠ ε, απορροφάται από τις άμεσες πληρωμές. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε το ερώτημα. Είναι οι άμεσες πληρωμές ο καλύτερος τρόπος στήριξης των παραγωγών. Τους βοηθάει να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά. Παραδείγματο χάρη, οι άμεσες πληρωμές αυξάνουν ή μειώνουν την κινητικότητα και την ε, επέκταση, την, ε, ανάπτυξη των ε, παραγωγικών μονάδων. Ορισμένες άμεσες πληρωμές βοηθούν και βελτιώνουν αυτούς τους στόχους, άλλες όμως όχι και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό πολύ προσεκτικά. Επίσης, βασικές πληρωμές και πράσινες πληρωμές. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι δύο τύποι πληρωμών δεν βελτιώνουν την παραγωγικότητα. Όμως, την πρόταση Υπάρχουν και άλλες προτάσεις που απευθύνονται ακριβώς σε αυτό το θέμα. Το ε, Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Προσαρμογής και τα μέτρα στον δεύτερο πυλώνα για την ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης ε, στα πλαίσια της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Εγώ πιστεύω κατά την εκτίμησή μου ότι οι δημοσιονομικές ε, παροχές ε, βάσει των νέων θεσμικών οργάνων είναι ανεπαρκείς. και χρειαζόμαστε νέα θεσμικά όργανα τα οποία άμεσα θα υποστηρίξουν και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα προκύπτουν ε, ναι, χρειαζόμαστε νέα θεσμικά μέτρα, διότι πιστεύω ότι οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν δεν συμβάλλουν όσο θα έπρεπε στην ανίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της έρευνας και τεχνολογίας ε, και της επίλυσης των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Νανία. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκίγιο Οι euh, διαφάνειες είναι στα αγγλικά, αλλά θα μιλήσω γαλλικά. Euh, το πρώτο μέρος αφορά αυτά το οποίο είπε ο κύριος Ανωνίας, γι' αυτό θα προσθέσω μόνο κάποιες παρατηρήσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την διατροφική ασφάλεια, διότι σήμερα πρέπει να παρέχουμε ήδη διατροφή σε 9 δις σε 7 δις, ενώ το 2050 σε 9 δις και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα προβλήματα, τα περιβαλλοντικά, τα ενεργειακά και νομίζω ότι η άνοδος των ανισοτήτων, των οικονομικών, των κοινωνικών και άλλων στις διάφορες χώρες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεύτερο σημείο, έχουμε να κάνουμε με μία ποσοτική πρόκληση, δεδομένου ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη ε, περισσότερο ένα δις μέχρι το 2050 και άλλο ένα δις ένα ε, δις υποσυτίζεται και ένα δις υπερσυτίζεται και είναι παχύσαρκο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να παίξουμε αν θέλετε σε θέματα κατανάλωσης και εδώ έχει σημαντικό ρόλο και η ΚΑΠ. Το πρώτος μας στόχος είναι να μειώσουμε τη φτώχεια. Δεύτερον, να μειώσουμε τις απώλειες και τις ε, διασπάθηση ειδών διατροφή και πώς θα μπορέσουμε να παρέχουμε στα διάφορα νοικοκυριά ε, φτωχά ή λιγότερο ε, ή περισσότερο πλούσια μια ισορροπημένη διατροφή. Ξέρουμε ότι αυξάνοντας την παραγωγικότητα θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο κάποια νεομοιογένεια και κάποιε ανισορροπίε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε σε επίπεδο γεωργίας να κάνουμε μία αηφόρο εντατικοποίηση και μία ισορροπημένη εναντικοποίηση παραγωγή. Δηλαδή να συνδυάσουμε την παραγωγή με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά τα λέγω για να δείξουμε πόσο ε, η αύξηση της ε, ανταγωνιστικότητα επηρέασε τα πράγματα σε σχέση με τι προηγούμενε δεκαετίε. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και θέλω να τα ναι. πάρουμε υπόψη. Ακόμη και στα πιο αισιόδοξα σενάρια, έχετε πολύ σημαντική αύξηση τη κανονική παραγωγή στι αναπτυσσόμενε χώρε και κυρίω στι χώρε τα πιο, πιο φτωχέ του κόσμου. Το 2030-40 θα πρέπει να γίνονται περισσότερε ανταλλαγέ γεωργικέ, ώστε να έχουμε εξαγωγικέ περιοχέ στην νότιο ε, την νότια παραγωγή και τη Ρωσία προ την Ασία, την υποσαχάρια περιοχή και την νοτιοανατολική Ασία. Ένα από τα σημαντικά θέματα λοιπόν σε αυτό το νέο σύστημα ανταλλαγών που βρίσκεται η Ευρώπη. Επίση, πολύ καλό νέο αυτό για του αγωγού. Θα πρέπει τα, τα επόμενα χρόνια θα δούμε ότι θα αυξηθούν οι τιμέ, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει σε επίπεδο παγκόσμιο. Θα υπάρχουν μεγάλε διακοιμάσει τιμών. Αυτό είναι καινούριο και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και μερικά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως ως στοιχείο να το λάβουμε υπόψη. Ε, δηλαδή, σχετικότητα του κόστους, διακοιμάσεις του κόστους, γιατί ε, λιγότερη προστασία στα σύνορα, κλιματικές αλλαγές και σχέση μεταξύ της τιμής τη ενέργειας και της τιμής των αγροτικών προϊόντων. Το βλέπετε εδώ δεξιά στη γραφική παράσταση και βλέπετε ποια είναι η τιμή του ε, πετρελαίου και ποια είναι η τιμή και η εξέλιξη της τιμής του καλαμποκιού. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όταν είναι οι τιμές αρκετά χαμηλές, δεν υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ των δύο, αλλά όταν υπάρχει αυξητική τάση υπάρχουν μεγάλες πιέσεις. Δεύτερο στοιχείο, σε επίπεδο κόσμου, όπως και σε επίπεδο Ευρώπης, υπάρχει ανάγκη να έχουμε έναν αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος να είναι παραγωγικός, ανταγωνιστικός, αηφόρος και ξέρουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις, τουλάχιστον στην Ευρώπη του βρεβάζουν από την άσκηση της γεωργίας που είναι αρνητικά, από το 2012 και μετά με τη μεταρρύθμιση της γεωργίας μειώνονται οι ε, αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά βεβαίως η αποδέσμευση ε, η οποία ακολουθείται δεν επαρκεί για να βελτιωθούν τα οικοσυστήματα. Και που καταλήγουμε, στα πλαίσια της ΚΑΠ θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποια κριτήρια, να έχουμε μέτρα στο δεύτερο πυλώνα, να βελτιώσουμε τα μέτρα του πρώτου πυλώνα, δηλαδή να προσέξουμε ακόμη περισσότερο τον, ε, τις προσπάθειες που κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Για να μπορέσει ο η φροντίδα προς το περιβάλλον να γίνει πραγματικότητα, θα πρέπει να δούμε πραγματιστικά τι συμβαίνει. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόοδο και η πρόοδος είναι ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε μέσα και σε μεθόδους οι οποίες ε, θα σέβονται το περιβάλλον. Υπάρχει επίσης το θέμα της διατροφικής ασφάλειας, της, ε, ε, των διακοιμάσεων του κόσμου και της αντιγωνιστικότητας. Δεν θα επανέλθω στην αηφορία και στην σταθεροποίηση. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στην πρόταση, στην νομοθετική πρόταση προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά βεβαίως θα πρέπει να γίνει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση τους, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τον κοινοτικό προπολογισμό και τα κονδύλια που θα δοθούν στην ΚΑΠ για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νέα πολιτική. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε με την αντιγωνιστικότητα. Αυτά τα λέγω για να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη ε, διακύμανση όσον αφορά τα εισοδήματα των γεωργών και ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα θέματα υπόψη. Τελευταίο σημείο σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα και την ΚΑΠ, και εδώ τελειώνω. Το πρώτο θέμα είναι, έχουμε θέμα ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια όλης της αλυσίδας της αγροδιατροφικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν μπορούμε να συνοψίσουμε σε ένα διάγραμμα το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την γεωργική παραγωγή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει στασιμότητα της παραγωγής στις αναπτυγμένες χώρες μετά από τον γύρο της Ουρουγουάης και τις διάφορες συμφωνίες που θεσπίστηκαν και υπάρχει μείωση των ε, επιδοτήσεων και βοηθειών. Απ' την άλλη βλέπουμε αύξηση της παραγωγής σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες και στις αναδυόμενες χώρες. Παίρνω τους αριθμούς ε, της ε, Βραζιλίας. Εδώ έχουμε αύξηση όσον αφορά την παραγωγικότητα. Εάν συγκρίνετε τι έγινε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, οι προτιμές παραγωγικότητα δεν βελτιώνεται εδώ, ενώ αντιθέτω βελτιώνεται στη ΣΥΠΑ. Άρα έχουμε διαφοροποίηση. Απ' την άλλη, η αύξηση ε, ανταγωνιστικότητας δεν έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, κυρίως για όποιες χώρες όπως η Γαρία. Και με εξαίρεση στη Γερμανία και κάποιες ε, για κάποιες άλλες νέες χώρες βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στον ισολογισμό. Αναλύουμε το, πρόγραμμα αυτό, το πρόβλημα αυτό για να δούμε κατά πόσον οι νέε προτάσει θα μα επιτρέψουν να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Και πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να απομονώσει κανεί ε, τον ε, ε, γεωργικό τομέα, τον αγροδιατροφικό. Θα πρέπει η προσέγγιση να είναι σφαιρική από το α μέχρι το ω της αλυσίδας. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με ένα διακύβημα σε σχέση με το τι παράγουμε εμείς σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι θέμα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το εσωτερικό πρόβλημα και τις ανοσορροπίες που υπάρχουν εντός των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη παρατήρηση. Εάν έχετε παραγωγικότητα και απόδοση μικρότερη σε κάποιες χώρες ευρωπαϊκές και συγχρόνως πρέπει να λύσετε και το πρόβλημα του ε, περιβάλλοντος, σε αυτά τα πλαίσια η πρωτοβουλία να εστιαστεί στούμε στα πλαίσια των προτάσεων στην καινοτομία είναι ένα καλό θετικό μέτρο και για να υπάρχει στα πλαίσια της παραγωγής και της αηφορίας συνεργασία θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να δούμε στα πλαίσια των πρωτοβουλίων που λαμβάνονται και που καταλήγουμε ότι θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πορίσματα της ε, βασικής έρευνας διότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, είναι θέμα γνώσεων. Ένα παράδειγμα. Σε θέματα γενομάτων, δηλαδή σε θέματα γονιδίων και έκφρασης των χαρακτήρων. Στα επόμενα δέκα χρόνια θα έχουμε να κάνουμε με μια πραγματική ε, ε, επανάσταση. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε τη σωστή έρευνα και ολοκληρωμένη και βασική για να μπορέσουμε να δούμε πώς όλα αυτά τα θέματα θα μπορέσουμε να τα ελέγχουμε αν θέλετε ή να τα γνωρίζουμε σωστά στα πλαίσια όλα της διατροφικής αλυσίδας. Τώρα όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πρόκληση και για μας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε μια κοινή αγορά για τα ΚΑΠ, αλλά όχι για τους διάφορες παράγοντες και τις διάφορες συνιστώσεις που συνθέτουν την γεωργία. Υπάρχουν εξηγήσει, όπως Φερρυπίν, έχουμε στασιμότητα της παραγωγής, αλλά το κόστος και οι υπόλοιπε συνιστώσεις δεν ε, μπόρεσαν να προσαρμοστούν έγκαιρα σε αυτή την κατάσταση. Δεύτερο, η συνιστόσα εργασία είναι ανομοιογενής μεταξύ των κρατών μελών και αν υπάρξει μείωση αυτής της συνιστώσης για την ΚΑΠ δεν είναι κάτι το βιώσιμο ως λύση μακροπρόθεσμα. Υπάρχει το θέμα του περιβάλλοντος που επίσης επηρέασε το κόστος παραγωγής περισσότερο όσον αφορά την κτηνοτροφία παρά τη γεωργία. Αλλά είναι αναγκαίο αυτό σε σχέση με την εναντικοποίηση την οικολογική και νομίζω ότι αυτό επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μην εστιαστούμε υπερβολικά στο κόστος, αλλά να λάβουμε υπόψη και την ανομοιογένεια των ε, γεωργικών ε, δομών και τα χαρακτηριστικά όλης της αγροδιατροφικής ε, αλυσίδας. Το μοντέλο της Ευρώπης όντως είναι ένα επικοινόμορφο μοντέλο, είναι αυτό ένα πλεονέκτημα, δηλαδή ρωτώ με εάν κάποια στιγμή αυτό δεν έχει σχέση και με μία έλλειψη εξειδίκευτη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ακόμα όμως δεν έχουμε επαρκή απαντήσει για το θέμα αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει υπερβολική υπερηφάνεια για το ευρωπαϊκό διατροφικό και γεωργικό μοντέλο. Και για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν περί τίνος πρόκειται οι καταναλωτές στην Ευρώπη θα κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια ε, ώστε να το μάθουν όλοι καλύτερα και να έχουν όλοι υπόψη τους την ποιότητα. Το θέμα που πρέπει να τεθεί είναι η ενίσχυση που θέλουμε να κάνουμε όλου του τομέα δεν θα είναι αντίθετη προς τον στόχο που θέλουμε να μην έχουμε περιθωποιημένες χώρες και οικονομία. Πιστεύω. Επίσης θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για την ικανότητα που θα έχουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση και να έχουμε υπόψη μα ότι κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε με πνεύμα αισιοδοξία. Τώρα, όσον αφορά την διαφοροποίηση των εισοδημάτων των ε, νοικοκυριών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εκτό από τι διάφορε διαστηριότητες που μπορεί να κάνει στο αγρόκτημά του, αυτό το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να μελετάμε, πράγμα το οποίο ακόμη δεν λαμβάνεται παρκώ υπόψη στις προτάσεις μεταρρύθμισης τη ΚΑΠ, είναι για να μπορέσουν να ε, διαποροφηθούν τα ε, εισοδήματα των γεωργών να συμπεριβλάβουμε και θέματα που αφορούν υπηρεσίες, υπηρεσίες, δηλαδή βελτίωση των υπηρεσιών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε αυτά από τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αναλάβουν οι γεωργοί σε κάποιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τα εισοδήματά τους. Ευχαριστώ. Oh, ε, Παρακαλώ τώρα να είναι πραγματικέ ερωτήσει που θα απευθύνεται, Αυθεντικέ ερωτήσει και όχι σχόλια και παρατηρήσει, διότι αλλιώ θα ξεπεράσουμε αυτή, αυτή τη, τη μισή που έχουμε στη διάθεσή μα για αυτό το κομμάτι τη συνάντηση. Έχει το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον πρόεδρό μας, τον επίτροπο και όλους τους προλαλήσαντες καθηγητές και εμπειρογνώμονες. Έχω ερωτήσεις και προς τους δύο καθηγητές. Μιλήσαμε για επισητιστική διατροφική ασφάλεια. Δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις στην Ευρώπη, τις οποίες λάβατε υπόψη. Ότι δηλαδή ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, αντί να παράγουν τρόφιμα, παράγουν ενέργεια και υποστηρίζονται οικονομικά. Η Βραζιλία κυβέρνηση πρόσφατα αποφάσισε εκατομμύρια εκτάρια να διατεθούν ε, για μία αγροτική παραγωγή. Ο Επίτροπος κ. Σιόλος ε, προτείνει ορισμένες αγροτικές εκτάσεις να βγουν εκτός παραγωγής. Είναι αυτή μία ε, ε, λογική πρόταση. Θα βοηθήσει στην επιστημιστική ασφάλεια ή θα βλάψει. Επίσης είπατε ότι αρκετά τρόφιμα ε, παράγονται εάν υπήρχε ισότιμη κατανομή. Όμως πρέπει να έχουμε τον ορίζοντά μας τραμμένο προς το 2050. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα αυξηθεί και άλλο ο πληθυσμός της γης, άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθεί και η αγροτική παραγωγή. Και τρίτον, εγώ πιστεύω ότι οι έρευνες πρέπει να υποστηριχθούν, να έχουν μία ισχυρή στήριξη. Όμως στη Γερμανία οι μικρομεσαίοι ε, κατασκευαστές αγροτικών μηχανημάτων μου είπαν ότι σε, στο Καλαμπόκι, παραδείγματο χάρη, 20 εκατοστά ε, στο αυλάκι καλλιεργούνται με σπόρους και το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα 50 εκατοστά δεν ε, φυτεύονται με σπόρους. Πώς λοιπόν μπορούμε να αυξήσουμε καλύτερα τα μηχανήματα, τα αγροτικά τα οποία ε, χρειάζονται, πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε καλύτερα και εγώ θα ήθελα να θέσω ορισμένες ερωτήσεις. Και οι δύο ε, ομιλητές είπαν ότι δεν έχει αυξηθεί η απόδοση, η αγροτική απόδοξη, διότι δεν έχουμε ενισχύσει όσο θα έπρεπε η έρευνα. Ε, μήπως όμως αυτό συμβαίνει διότι έχουμε πλέον εκμεταλλευτεί τόσο πολύ τη γη και τα και τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα, ώστε να μην μπορούμε να αυξήσουμε πλέον την εκμετάλλευσή του. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο, στο όριο της εκμετάλλευσης. Έχει κορεστεί η εκμετάλλευση. Επίσης, δεν ακριβένουν συνεχώς τα μέσα παραγωγής. Ίσως και αυτό είναι ένα πρόσκομα στην αύξηση της παραγωγής. Η υπερεκμετάλλευση των πρώτων πόρων και των πρώτων υλών και ε, πολύ ακριβό κόστος παραγωγής αναφέρατε την αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρώπη. Ε, ασφαλώς θα έχετε σημειώσει ότι εισάγουμε όλο και περισσότερα αγροτικά προϊόντα, παραδείγματο χάρη σόγια ε, για ζωοτροφές, αλλά ε, κάνουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλες εισαγωγές. Και αυτό έχει επιπτώσει στην κρεατοπαραγωγή, στο κόστος δηλαδή ε, μελετώντας και συζητώντας αυτά τα θέματα παράλληλα με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και με τους ε, ενδιαφερόμενους του τομέα, ε, κατάλαβα ότι παρόμοιες συζητήσεις θα γίνουν και στα πλαίσια του Μερκοσούρ. Και επειδή υπάρχουν περιφέρειες στον κόσμο ε, και πολυμερείς συμφωνίες οι οποίες είναι επιτυχείς, υπάρχει ο κίνδυνος να παραγκονιστεί η Ευρώπη. Ε, είπατε ότι χρειαζόμαστε μέχρι το 2050 μία αύξηση του 70%. Είναι αυτό επίσημο στοιχείο του ΦΑΟ. Εγώ δεν έχω ακούσει αυτά τα στοιχεία ε, και δεν έχω ακούσει ποτέ το ΦΑΟ να ζητήσει 70% αύξηση της αγροτικής παραγωγής μέχρι το 2050. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστο αυτό το στοιχείο και από πού προέρχεται. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, για την ανταγωνιστικότητα. Ομως θα πρέπει να βελτιωθεί και άρα να αυξηθεί η παραγωγή. Σήμερα βλέπουμε ότι από τότε που ξεκίνησε η ΚΑΠ έχουμε τόση αύξηση παραγωγής όσο είναι και η διασπάθηση στην διατροφική αλυσίδα. Επομένως, αυτό είναι το θέμα πόσο έχουμε κερδίσει από τη μια πλευρά και έχουμε χάσει από την άλλη. Επομένως αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που είπατε και παρακαλώ πέστε μας δύο λόγια παραπάνω. Δεν λέει τίποτα το να παράγουμε περισσότερο εάν διασπαθίζουμε περισσότερο όσον αφορά την ε, ζωική παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο. Τι θα γίνει όσον αφορά την αλλαγή του διατροφικού προτύπου του διατροφικού μοντέλου. Αυτό είναι ένα πραγματικά σοβαρό ερώτημα σήμερα, γιατί έχουμε μια μεριά την κλιματική αλλαγή, την υπερθέρμανση και από την άλλη μεριά θα πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα της πρωτεΐνης ανά πρόσωπο. Και επομένως όμως λένε ότι η όξη παραγωγής ε, αυτό δεν αρκεί γιατί χρειάζονται πάρα πολλές ε, φυτικές πρωτεΐνες για να παραγάγουμε τις ε, ζωικές πρωτεΐνες. Τώρα επίσης όσον αφορά την αηφορία, την βιωσιμότητα υπάρχει κάτι το οποίο δεν το άκουσα ακόμα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο όμως μπορείτε να μας μιλήσετε. Δηλαδή τι γίνεται όσον αφορά τους φυσικούς πόρους που στηρίζουν την ε, ε, ζωική παραγωγή. Ποτάσιο, ε, φωσφορούχα, εκεί πέρα και εκεί είναι, είναι πεπερασμένοι οι, οι πόροι. Ισχύει αυτό. Και αν ισχύει τότε είναι πραγματικό πρόβλημα. Άρα τι, τι μοντέλο γεωργικό θα έχουμε. Διαβέστε μας γι' αυτά όσον αφορά λοιπόν την αλλαγή των μεθόδων παραγωγής σε σχέση με, τη, την Ευχαριστώ λέει πρόεδρος νόση. Έχουμε Ευχαριστώ Όλο και περισσότερο στην Ευρώπη βλέπουμε ότι παράγεται ενέργεια από, τις από την καλλιεργήσιμους ε, και όχι αγροτικά προϊόντα. Και οι πραγματογνώμονες μας λέγουν ότι με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι τιμές των αγροδιατροφικών προϊόντων. Βλέπουμε σύντομα αύξηση 7% στην τιμή αυτής της ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξηθούν και οι τιμές των ειδών διατροφής. Και όχι μόνο αύξηση των τιμών θα προκαλέσει αυτή η κατάσταση, αλλά και εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών μια κάποια ακαταστασία όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Για τα δημητριακά καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και πόσο η αγορά των δημητριακών ε, επηρεάζει και τα υπόλοιπα αγροτικά τρόφιμα. Θα πρέπει να βρούμε και ένα σύστημα αποθήκευσης των ε, δημητριακών για να μην φτάσουμε σε κατάσταση ελλημάτων. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Στην Ευρώπη έχουμε όλο και λιγότερο καλλιεργήσιμες γέες. Στην Πολωνία το 2007 το Ευρωμαρόμετρο μίλησε για 16 εκατομμύρια εκτάρια περίπου. Σήμερα έχουμε 15 εκατομμύρια. Και ακόμη λιγότερες ε, ε, επιφάνειες ε, οι οποίες επιδοτούνται. Αρρώσιμες οι οποίες επιδοτούνται. Αυτό δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα και άλλων χωρών. Βλέπουμε ότι η μείωση αυτή αυξάνεται εκεί που υπάρχουν λιγότερες επιδοτήσεις ανά εκτάριο. Και το αντίθετο συμβαίνει εκεί που δεν υπάρχουν. Υπάρχει άμεση σχέση. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη, κύριε εμπειρογνώμονες. Δηλαδή, ότι πολύ μικρές επιδοτήσεις ανά σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης σημαίνει ότι έχουμε λιγότερες ε, αρρώσιμες επιφάνειες διαθέσιμες, πράγμα το οποίο θέτει εν κινδύνο τη διατροφική μας ασφάλεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους, το πάνελ και όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα να επανέλθω σε μια παρατήρηση που έγινε ότι πρέπει να συνδυάσουμε την παραγωγή και το περιβάλλον. Γιατί πρέπει να το πούμε τώρα αυτό και πού, κάναμε τόσα μεγάλα λάθη και γιατί. Ε, ποια ήταν τα μεγάλα μας λάθη ώστε τώρα να προσπαθούμε πάλι να συνδυάσουμε κάτι το οποίο είναι προφανές από παλιά. Δεύτερον, όσον αφορά τώρα τη χρήση της γης, ε, ε, ε, έχω κάπως μπερδευτεί το να συνδυαστεί ε, η ιδιοκτησία ε, ή η καλλιέργεια διαφόρων ε, φυτών ή η αγρανάπαυση. Δηλαδή το να μοιράσουμε τη γη ή να την βγάλουμε εκτός αγροτικής παραγωγής. Επίσης, αν δείτε την παγκόσμια κατάσταση, προσπαθούμε να ανταγωνιστεί η Ευρωπαϊκή Γεωργία της. Ε, τους αγροτικούς τομείς ολόκληρης της συμφιλίου. Πώς μετράτε την ανταγωνιστικότητα με τέτοιες ε, συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή ε, τι άλλα μετρήσιμα ορόσημα έχετε για να πείτε ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι ανταγωνιστική ή δεν είναι και πόσο είναι ανταγωνιστική έναντι των άλλων. Μπορείτε να σχολιάσετε τις πληρωμές του πυλώνα 1 που κυρίως αφορούν ε, ε, το εισόδημα και εδαφικές, εδαφικά κριτήρια. Πιστεύετε ότι οι πληρωμές αυτές είναι θετικές του πρώτου πυλώνα. Ευχαριστώ κύριε. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε το κατάλληλο των αγορητών. Ε, άλλοι τρεις έχουν το λόγο, αλλά προς, προσοχή να μείνει πιο πρόσφατο χρόνο μας. Καπούλιας, Άγνιου και κατόπιν κάποιος άλλος έχει το λόγο. Λουίς. Λουίς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Πίτρο και τον κύριο Υπουργό γιατί είναι παρόντες και να ευχαριστήσω όλα τα άτομα που είναι εδώ. Απλή ερώτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις ναι, έκθεση της κατάστασης της ΚΑΠ που έκαναν οι δύο ε, εμπειρογνώμες. Κάναν πάρα πολύ ανάλυση, επικριτική, αλλά λείπει κάτι το οποίο προσδοκούσαμε εμεί περισσότερο. Ποιε είναι οι λύσεις που προτείνονται. Ο καθηγητής κ. Ανανία είπε ότι βρίσκονται προς την καλή κατεύθυνση οι προτάσει, αλλά τα μέσα που προτείνουν είναι ανεπαρκή. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία είναι ανεπαρκή και τα οποία λείπουν για την άποψή σα. Ο κύριος Γκίγιομάρ είπε ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη οργάνωση επιτροφή και μία ε, και πολύ περισσότερες προτάσεις και λύσεις. Οι αποφάσεις είναι θέμα πολιτικών. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε εμείς βάσει των στοιχείων που μας δίνουν οι επιστήμονες τι λύσεις θα προτείνουμε και τι αποφάσεις θα πάρουμε. Περιμέναμε μεγαλύτερη βοήθεια από τους επιστήμονες. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποιες είναι οι αποτελεσματικές κατά την άποψή σας και οι πραγματικές ε, ελλείψεις που επισημαίνετε και μπορείτε να μας κάνετε κάποιες προτάσεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τρεις ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι η απόρριψη αλλιευμάτων ε, στο βυθό της θάλασσας είναι παραγωγικός τρόπος χειρισμού της γεωργίας, δεν θα μπορούσαν αυτά να χρησιμοποιηθούν ως τροφές. Επίσης, ε, τα απορρίμματα γενικά των σφαγείων χρησιμοποιούνται κατά πολύ κακό τρόπο και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον ορισμένα κομμάτια σαν, ως λείπασμα. Ε, δεν μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω το κόστος παραγωγής χρησιμοποιώντας ε, χρήσιμα στοιχεία των αποβλήτων και απορριμμάτων. Ακόμη ένα άτομο είστε στο λόγο, πείτε μας το όνομά σας. Ναι, γεια σας. Είμαι ο Πέντρο Νάρο, εκπρόσωπο την, ε, Νασάχα, τους αγρότες Τη Ισπανίας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μιλήσατε για ανταγωνισμό και το ερώτημά μου είναι πρέπει να παράγουμε περισσότερο, πρέπει να μιλάμε για καλύτερη διαχείριση των πόρων. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να σας διαφεύγει ο τρίτο πυλώντα, τα εισοδήματα των γεωργών. Θα πρέπει να προσπαθήσετε τα δίκαια εισοδήματα των γεωργών να τα διασφαλίσετε, διότι αν συνεχίζουν να πουλούν σε τιμή κάτω του κόστε, δύσκολο θα μπορέσετε να εφαρμόσετε τι νέε τεχνολογίε και την καινοτομία. Συγκεκριμένα, για να είμαστε πιο αντιγωνιστικοί και να είναι οι αγρότε πιο ανταγωνιστικοί. Κυρία Νανία, τι είδου προτάσει ειδικέ θα κάνατε εσεί ώστε στα πλαίσια τη μεταρρύθμισης της ΚΑΠ να μπορέσει να υπάρξει εξισορρόπηση των ε, δύναμη των αγροτών και των άλλων μετεχόντων στην διατροφική αλυσίδα. Επίσης, είπατε ότι η πράσινη πληρωμή, αν θέλετε, και η δίκαια πληρωμή δεν είναι πολλές φορές ε, η κατάλληλη λύση για τον ανταγωνισμό. Όπως είπε και ο κύριος Καπούγιας, πείτε μας κάποια μέτρα. Πώς μπορούμε εμείς ε, να αλλάξουμε τα πράγματα όσον αφορά την πράσινη πληρωμή για να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Τρίτον, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καινοτομία και ε, για ανταγωνισμό εάν αρνούμεθα την πράσινη βιοτεχνολογία να την εφαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, καθηγητής κύριος Ανανία και ο καθηγητής κύριος Γκίγιο Μάρ έχουν το λόγο για να απαντήσουν. Uh, Αναρωτιέμαι πόσο ε, χρόνο έχουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα πολύ κέρια ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όσον αφορά την ενέργεια, αποφάσισα στο, στα 10 λεπτά χρόνο μιλία που είχα να μην μιλήσω για την ενεργειακή πολιτική και τα βιοκαύσιμα. Αλλά όταν μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο για διατροφική ασφάλεια, Ασφαλώς, η πιο σημαντική πολιτική που έχει επίπτωση στην διατροφική ασφάλεια είναι η πολιτική μας για τα βιοκαύσιμα. Η πολιτική μας για τα βιοκαύσιμα είχε βεβαίως ως αποτέλεσμα τη μείωση της αγροτικής παραγωγής και την αύξηση του κόστους. From uh, security. Όσον αφορά τώρα την πτυχή της διατροφικής ασφάλειας, πρέπει να βελτιώσουμε την πολιτική μας για τα βιοκαύσιμα και την, την, ε, τις εμπορικές, την εμπορική μας πολιτική για τα βιοκαύσιμα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές αυτής της ε, ιδιαίτερης πολιτικής. Και αυτό που πρέπει επίσης να μελετήσουμε είναι τη σημασία της έρευνας και ανάπτυξης ε, το, για τα βιοκαύσιμα από ενεργειακής πλευράς αν ε, αναπτύξουμε την έρευνα και τεχνολογία θα καταλήξουμε ελπίζω στη χρήση λιγότερης ενέργειας και θα βρούμε τρόπους πιο επικοδομητικούς και πιο αποτελεσματικούς στην παραγωγή των βιοκαυσίμων. Ε, πρέπει να μειωθεί η επίπτωση των, της παραγωγής βιοκαυσίμων στην επισητιστική ασφάλεια η διασύνδεση μεταξύ επενδύσεων ε, ε, για την έρευνα και τεχνολογία και των αλλαγών στην παραγωγικότητα. Οι εμπειρογνώμονες μου έχουν πει ότι υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει εύρος να, να, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Ε, εάν βελτιωθούν οι πολιτικές που εφαρμόζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως οι επενδύσεις στην ανάπτυξη και την έρευνα δεν ε, θα έχουν ε, αποτέλεσμα μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά θα φέρουν αποτελέσματα και στις ε, περιβαλλοντικές πτυχές της αγροτικής παραγωγής. Έρευνα και ανάπτυξη λοιπόν και για περιβαλλοντικούς σκοπούς. Ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα Κάταρχα δεν σημαίνει ότι πρέπει το μόνο στοιχείο στο οποίο οφείλεται είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Υπάρχουν αγροτικά συστήματα που λειτουργούν στην Ευρώπη και ο τρόπος για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα δεν είναι τόσο πολύ μείωση του κόστου παραγωγής, αλλά στην αύξηση ε, της ποιότητας των προϊόντων, δηλαδή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και ενώ βελτίωση της ποιότητας τι εννοώ, εννοώ όλα τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία ζητάνε οι καταναλωτές και υπάρχουν πολλές διαφορετικές δέσμες ποιοτικών ε, κριτηρίων, ποιοτικών προδιαγραφών. Παραδείγματος χάρη, η βελτίωση των, της ε, ευημερίας, ευζοίας των ζώων ε, από, να ας ξεκινήσουμε από εκεί μέχρι τις ε, καμιά φορά ε, πάρα πολύ ψηλέ απαιτήσει των πλουσίων καταναλωτών. Μέσα στην γάμα αυτή των ποιοτικών κριτηρίων πολλά μπορούμε να βελτιώσουμε. αυτό που θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγικότητας. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις μεθόδους παραγωγής ανάλογα με ε, τις παραγωγικές μονάδες, με τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Δεν είναι δυνατόν όλα τα αγροτικά συστήματα να τα βάλουμε σε, μία πλατφόρμα και να πούμε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Όλα τα ε, παραγωγικά συστήματα στις μονάδες πρέπει να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για να ακολουθούν τα δικά τους κατάλληλα μέτρα. Γι' αυτό πρέπει να καθορίσουμε το, τα στοιχεία αυτά της ΚΑΠ τα οποία χρειάζονται μεταρρύθμιση. Παραδείγματο χάρη, να βρούμε τρόπους να μην φεύγουν οι νέοι ε, παραγωγοί, τα παιδιά των αγροτών από τις ε, παραγωγικές μονάδες, να μην εγκαταλείπουν την ύπεθρο και τέτοια μέτρα λοιπόν. Τώρα, ο δεύτερος πυλώνας, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκεί και τι γίνεται με τον πρώτο πυλώνα για μένα, επειδή πιστεύω ότι έγινε αναφορά σε διπλές ε, ε, πληρωμές, διασυνδεδεμένες πληρωμές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τις άμεσες πληρωμές δεν είναι αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά ενίσχυση της υπαίθρου, ενίσχυση της αηφορίας, της, ε, του αγροτικού τομέα, και διαμόρφωση των συνθήκων της αγοράς έτσι ώστε να μπορεί να επιζήσει η γεωργία και η αγροτική παραγωγή σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Ε, Τώρα έχουμε και ορισμένες εύκολες ερωτήσεις, αλλά οι απαντήσεις είναι δύσκολες. Αυτό συνήθως συμβαίνει. Ε, η ακαδημαϊκή κοινότητα λέ, μας λένε συχνά ότι ωραία μας τα λέτε, αλλά τι θα κάνετε εσείς στη θέση μας, αν κάνατε εσείς τη δουλειά μας. Η άποψή μου για την μεταρρύθμιση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής είναι ότι δεν επαρκούν οι προτάσεις. Δεν είναι αρκετά ριζικές και ε, ε, επαρκείς. Πολλά, που πολλά μέτρα που προτείνονται στη μεταρρύθμιση in sustainable and effective way and Πολλά μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα είναι καλά για τους νέους παραγωγούς και θα τους επιτρέψουν να είναι πιο ανταγωνιστικοί, να επιβιώσουν, να βελτιώσουν το εισόδημά τους κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι άμεσες πληρωμές κατά ένα ποσοστό για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε στοχευμένα μέτρα τα, τα οποία θα βοηθούν την ποιότητα, θα βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και γι' αυτό πιστεύω ότι οι παρούσες προτάσεις δεν είναι τόσο ολοκληρωμένες και πλήρεις όσο θα ήθελα. Οι άμεσες πληρωμές θα πρέπει να έχουν ως στόχο να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής και την μείωση της ανταγωνιστικότητας. Δεν θα πρέπει ε, στα δημόσια αγαθά οι άμεσες πληρωμές να έχουν αυτή την, την ίδια αρνητική επίπτωση που έχουν στους παραγωγούς. Άρα πρέπει ορισμένους πόρους σιγά σιγά να τους βγάλουμε από τις άμεσες πληρωμές και να τους διοχετεύσουμε εκεί όπου χρειάζονται μέτρα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Διότι σε 20 χρόνια δεν θα πρέπει να λέμε πια τι θα κάνουμε με αυτές τις άμεσες πληρωμές οι οποίες συνεχώς φθήνουν, φθήνουν, φθήνουν, φθήνουν. Θα έπρεπε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Σταματώ εδώ και θα δώσω το λόγο στον Ερβέ. Να απαντήσει τα πιο δύσκολα. Σας ευχαριστώ. Προσπαθήσω να συμπληρώσω τα όσα απήντησε ο συνάδελφος Σαββατεμέρη να σας πω ότι αυτή η διατροφική πρόκληση η παγκόσμια δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε απομονωμένα από τις άλλες προκλήσεις που ταυτόχρονα αναδύονται. Είναι η ενεργειακή, όσον αφορά τα όρια, τα καύσιμα κλπ. Έχουμε το περιβάλλον σαν πρόκληση και τώρα έχουμε επίσης και τις ανισότητες. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε τις πολιτικές υπέρ των βιοκαυσίμων ας πούμε σε σχέση και όχι ενάντρια σε κάτι άλλο το οποίο βοηθάει την αγορά να αγκαλιάσει τη βιομάζα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τώρα τα βιοκαύσιμα που με τίποτα δεν είναι πανάκια αυτή η πρώτη γενιά από αυτά τα καύσιμα να συνεχίσουμε με τις προσπαθειές μας σε σχέση με τις άλλες γενιές από αυτά τα καύσιμα που θεωρείται ότι θα αποτελούν παράγοντα ανταγωνιστικό στην ε, διατροφική παραγωγή επίσης. Όσον αφορά τώρα της παραγωγικότητας και εδώ πέρα έχουμε πολλές ερωτήσεις ή στην Ευρώπη υπάρχει η δυσκολία η εξής. Έχουμε εδώ και τόσα χρόνια ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο πάρα πολύ καταπήγε. Τόσα χρόνια δηλαδή. Τελικά έγιναν κάποιες επιλογές για τα λοιπάσματα, Φερρυπίν. Τα λοιπάσματα τα οποία βοηθούσαν τη μεγαλύτερη παραγωγή το σύστημα αυτό στην αρχή ήταν συμπαγέ, αλλά σιγά σιγά φάνηκαν κάποια αρνητικά επί του περιβάλλοντος και άρα τώρα θα πρέπει να περάσουμε σε κάποια άλλα συστήματα. Πιο διαφοροποιημένα και πιο πολύ προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους του κάθε μέρους, κάθε τοποθεσία, όπω πούμε τα σχετικά με τα φυτο-υγειονομικά, ας πούμε για τα ζυζανιοκτώνα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ολοκληρωμένη παραγωγή και άρα θα πρέπει να συνδυαστούν διαφορετικές μεταβλητές. Και γι' αυτό και είναι σημαντικό να έχουμε συνεργασία όλων αυτών των εμπλεκομένων γεωργών, δημόσιου τομέα, ιδιωτικού τομέα, αναπτυξιακών φορέων και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσει η Ευρώπη έτσι να διατηρήσει την παραγωγικότητά τη αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Το οποίο πραγματικά όμως είναι δύσκολο, γιατί χρειάζεται τώρα να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο διαφοροποιημένη προσπάθεια. Τώρα, τι λύσεις έχουμε προτείνουμε. Τελικά θα καταφέρουμε να δούμε τι είναι πιο αποδοτικό, τι είναι πιο αποτελεσματικό σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Γιατί έχουμε τα σχετικά μέτρα απολυτικής να αναζητήσουμε και κάποιους διαφορετικούς πόρους τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, τις διαφορετικές ζώνες ανάπτυξης. Στο Μόναχο, ας λέμε τη σχετική περιοχή και θα πρέπει να προσπαθήσουμε τόσο ώστε να ξεπεράσουμε τα δημοσιονομικά όρια και δημοσιονομικούς περιορισμούς. Είμαστε πολύ πιο τολμηροί από ό,τι σήμερα, από ό,τι είναι σήμερα η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη. Και άρα, έτσι, βρίσκουμε και λύση όσον αφορά την παραγωγικότητα. Που είναι πάρα πολύ σημαντική για την επιβίωση της γεωργίας αλλά και της γεωργικής βιομηχανίας. Άρα δεν είναι θέμα μόνο μεγαλύτερης, περισσότερης παραγωγής. Θα πρέπει μόνος να υπάρξει ποικιλία στη δραστηριότητα, διαφοροποίηση πέραν της καθαρά παραγωγής διαδικασίας. La valeur ajoutée que vous pouvez distinguer, et là je pense aussi qu'il y a du travail à faire. Par rapport à... Τώρα, για να δούμε παρακάτω τι γίνεται όσον αφορά την ύπεθρο, τη γη στην Ευρώπη. Είπατε ότι δεν ήταν επαρκής οι ενισχύσεις και γι' αυτό και χάθηκε η γη. Ε, την άλλη μεριά εκεί που υπήρχαν σημαντικές ενισχύσεις, δεν καταλαβαίνω πώς το σχετίζει ένα με το άλλο. Ή έχουμε περίσευμα γης σε σχέση με το τι ζητάει η αγορά ή υπάρχει ζήτηση για άλλη χρήση παρά για τη γεωργία. Δεν δε φταίνε δηλαδή ενισχύσει σε σχέση με το ότι πάει η γη σε άλλες δόσεις από τη γεωργία. Άρα είναι θέμα τη εγκυοβελτιωτική της πολιτικής που ακολουθείται για τη γη. Θέμα κυριότητας, διαχείρισης της γης. Έτσι επομένω θα ζητηθεί θα συζητηθεί η λύση και όχι μέσω του τι θα κάνουμε με τις ενισχύσεις της επιδοτήσεις. Τώρα, τι θα γίνει με τα ηχθιάλευρα, αυτά τα, τα, οποία απορρίπτουμε, αυτά τα οποία λέει ο ΦΑΟ. Στο επίσημο website έχουν παρουσιαστεί κάποια στοιχεία Είναι επίσημα στοιχεία αυτά, αλλά από μόνα τους δεν λένε τίποτα. Όσο λιγότερο διασπαθίζετε, τόσο λιγότερο θα χρειάζεστε αύξηση της γεωργικής παραγωγής. Αυτό λέει το μήνυμα. Και εμείς, οι οικονομολόγοι, λέμε ότι έτσι μπορεί να υπάρξει κάποια απάντηση μέσω κάποιες ανάλυσης και γι' αυτό τώρα έτσι να δούμε πώς θα σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη διασπάθηση των πόρων το οποίο είναι δύσκολο. Δύσκολο γιατί θα πρέπει να ξεσυνηθίσουμε αυτές τις ανέσεις που δεν είμαστε έτοιμοι περισσότερο στην Ευρώπη να κάνουμε. Και υπάρχει μια βρετανική μελέτη πρόσφατη σε σχέση με αυτή τη διασπάθηση σε διανομή και κατανάλωση. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε 10% μείωση αυτής της διασπάθησης των πόρων. Άρα από εκεί θα καταλάβετε όπου έχουμε αυτή την προσπάθεια από το δημόσιο αλλά και από τα φυσικά πρόσωπα μέσω της παιδείας και τα παιδιά συμβάλλουν αλλά κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης ο κόσμος τώρα προσέχει περισσότερο. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα αυτή τη μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νανία και κύριε Γκυγιομάρ. Νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις σας τελειώσαμε τη σύντηση του πρώτου θέματος. Τώρα θα ήθελα να καλέσω την κυρία ε, Φρυμπάουερ γεωλόγο, λόγο από το Von Tunen Institute κλιματικών και ε, αγροτικών μελετών της μελέτης και τον καθηγητή Book Backwell. Καθηγητή γεωργικής οικονομίας του Imperial College του Λονδίνου για να μιλήσουμε για την αηφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως συνήθως, παρακαλώ τους παρεμβαίνοντες να προσπαθήσουν να μην ξεπεράσουν ο καθένας τα 10 λεπτά ώστε να έχουμε χρόνο για τις απαντήσεις μετά. Ευχαριστώ. So, so now, um, hello everybody. Yes. σας. In the next 10 minutes or so to um, Θέλω να, να προσπαθήσω τουλάχιστον να σας προτείνω ορισμένες λύσεις και να συνδυάσω το θέμα αυτό με περιβαλλοντικές διαστάσεις. Καταρχάς, ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Και καθώς οδεύουμε προς το 2020 αλλά και πέρα αυτής της ε, χρονολογίας. Ε, μιλάμε συνέχεια για την κλιματική αλλαγή και είναι σαφές πλέον ότι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι πιστεύουμε ακόμα πριν από δύο-τρία χρόνια. Έχουμε πλέον τώρα ε, πληροφορίες ε, αξιόπιστες που δείχνουν ότι η βιοπικιλότητα φθήνει, μειώνεται και το δύο, ε, ο στόχος μας η κλιματική αλλαγή να παραμείνει κάτω από δύο βαθμούς Κελσίου φαίνεται πλέον ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Επίσης ε, η ταχύτητα των αλλαγών αυξάνεται και στα, σε ευρωπαϊκή διάσταση η μεγάλη πρόκληση είναι να συμφιλιώσουμε την παραγωγή με την προμήθεια παρκών δημοσίων αγαθών. Ε, η απαραίτητη απάντηση την οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα εν ώψη των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της αλλαγής του κλίματος σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές και στην κατανάλωση και στην παραγωγή. Χρειαζόμαστε λοιπόν αντισταθμιστικά μέτρα για την, ε, για την αλλαγή αυτή του κλίματος και την διασφάλιση της βιοποικιλίας, της ποιότητας του νερού, των υδάτων και της ε, γης, του εδάφους. σε έναν κόσμο όπου η αστάθεια και το, τα, η κίνδυνη, το ρίσκο αυξάνεται συνέχεια, πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα ε, του ευρωπαϊκού συστήματος. Ε, όχι να βελτιώσουμε τη διαχείριση του ρίσκου, αλλά να ενισχύσουμε ε, συστημικά την πολιτική μας. Ε, τώρα η ερώτηση που βλέπετε εδώ είναι εάν η αηφορία ε, μπορεί να διασφαλιστεί με την ταχύτητα που χρειάζεται. Δυστυχώς, οι παρούσες προτάσεις για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, δεν, δεν έχουν λάβει υπόψη ένα, μια σταθερή πολιτική και σαφή πολιτική για τις ε, μελλοντικές αγροτικές και περιφερειακές περιοχές, τις περιφέρειες μάλλον, ε, και δεν είναι αρκετά φιλόδοξα αυτά τα μέτρα. Επίσης δεν ξεκαθαρίζουν πού πρέπει να βαδίσουμε και τι θέλουμε να επιτύχουμε. Ε, στο θέμα της αηφορίας πάντοτε. Αυτό επίσης λείπει είναι μια σαφής οικονομική πολιτική, δηλαδή πώς ο προπολογισμό να μπορεί να καλύψει ακριβώς τις απαιτήσει της αηφορίας. Θα επανέλθω όμως στα οικονομικά ε, λίγο αργότερα. Και τέλος, ε, δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο, έναν όγκο τεκμηρίωσης ε, οδηγιών, κανονισμών κτλ πρέπει να μην επιβαρύνουμε τα κράτη-μέλη με περισσότερα εμπόδια, αλλά να αφήσουμε να λειτουργούν κανονικά, τουλάχιστον στα θέματα αυτά στα οποία είναι επιτυχή. Δηλαδή, να εξακολουθήσουν την καθημερινή τους λειτουργία και εργασία. Δηλαδή, να είναι σαφές ότι τα θετικά στοιχεία πραγματικά χρησιμοποιούνται επικοδομητικά. Ποια, ποιοι είναι λοιπόν οι εφικτοί στόχοι για το 2020 όταν εννοώ εφικτά, εφικτούς στόχους, εννοώ τα ελάχιστα πρότυπα τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε με μέτρα τα οποία έχουν καθαρή στόχευση. Καταρχάς, ε, πρέπει να επιδιώξουμε μία επάρκεια πόρων και περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά. Πρέπει λοιπόν κατά 10 με 30% εάν μειώσουμε την ενέργεια και τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων κατά 10 με 30% δεν θα επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Δεν είναι επαρκή αυτά τα μέτρα. Επίσης πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη την την εδαφική διάβρωση πρέπει να βελτιώσουμε τη διαχείριση του εδάφου σε όλες τις ευάλωτες ζώνες. Ε, και θέλουμε επίσης να μειώσουμε την απώλεια της βιο, όπως ε, σας είπα, ορισμένα μέτρα για να αντισταθμίσουν αλλαγή κλίματος ε, είχαμε πει ότι θα ήταν 20% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην γεωργία και στη δασοπονία μέχρι το 2005 και προσαρμογή της, βιο... ποικιλία σε διάφορες περιφέρειες, ε, παραγωγικά συστήματα και μέσα σε παραγωγικές μονάδες. Αυτά τα είχαμε ήδη αποφασίσει και συζητήσει, αλλά τώρα είμαστε ενώπιση της μεταρρύθμισης. Για μένα ο πρώτος πυλώνας είναι ε, λίγο πολύ ε, απαράλλακτος. Δηλαδή δεν αλλάζει και τίποτα. Όπως λέμε στα αγγλικά, business as usual. Δηλαδή, ό,τι γινόταν πριν θα γίνει και τώρα ή και αργότερα. Το 75%, το 75 του budget, όπως είπαμε, χαραμίζεται στις ε, άμεσες πληρωμές. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μετρήσουμε αν αυτές οι άμεσες πληρωμές ποσοτικά αντισταθμίζονται με αντίστοιχα ωφέλη για τους παραγούς και δεν βρήκαμε αυτή την ποσοτική ε, σχέση ωφέλειας μεταξύ του όγκου των άμεσων πληρωμών και των ε, παραγωγικών ε, πλεονεκτημάτων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν αυτό. Η, όπως σας είπα, η κλιματική αλλαγή απαιτεί επάρκεια πόρων. και πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης αλλαγή της, εδαφικής, της ε, ιδιοκτησίας ε, της αγροτικής γης. Ε, μπορεί ένα αγροτικές εκτάσεις οι οποίες έμειναν ακαλλιέργητες ας πούμε μετά από μερικά χρόνια να ξανακαλλιεργηθούν. δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν η διατήρηση των παλαιών ε, λιβαδικών εκτάσεων είναι, καλό, είναι καλή για βιοπικιλία. Πρέπει να κλείσουμε ορισμένα παραθυράκια που υπάρχουν, όπως σας είπα, αλλαγή διοκτησίας και ε, πρέπει να βελτιώσουμε το οργανικό, ε, το οργανικό περιεχόμενο, το οργανικό ποσοστό, το ποσοστό οργανικών ισουσιών στο έδαφος για καλύτερη παραγωγή, πιο καλή ποιότητα. για να μπορέσουμε να συνδέσουμε καλύτερα, να συνδυάσουμε μάλλον καλύτερα την ε, παραγωγή ε, φυτών και εκτροφή ζώων με την ποιότητα του εδάφους. Κάθε περιφέρεια, όπως είπαμε, είναι διαφορετική και η δαπάνες οι οποίες σημειώνονται, οι δαπάνες οι οποίες συναπάγονται τα διάφορα μέτρα είναι διαφορετικά. Ε, άρα λοιπόν ε, οι άμεσες πληρωμές δεν μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους συνδυασμούς που θέλουμε. Ε, η, τύχη, η πρόταση λοιπόν είναι να, βελτιώσουμε, να μειώσουμε σταδιακά τις άμεσες πληρωμές. Ο δεύτερος πυλώνας τώρα είναι, περιέχει ορισμένες πάρα πολύ καλές αρχές ε, και ορισμένες ε, αρνητικές, ε, ορισμένα αρνητικά στοιχεία. Καλύπτει το απορροφά το 25% του συνολικού προϋπολογισμού. Και δεν μπορέσαμε να ανατρέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που, που σημειώθηκαν, ιδίως στη βιοποικιλότητα. Διότι ε, σημειώσαμε ότι πολλές φορές ε, δεν υπήρχε περιφερειακή συνοχή και συνέπεια στον προγραμματισμό των διαφορών πολιτικών. Οι εθνικές στρατηγικές τα στρατηγικά προγράμματα και η υλοποίησή τους είναι κρίσιμα για την αηφορία και ε, γι' αυτό ε, πρέπει να μειώσουμε ή να έχουμε ένα όρια όριο για τη συγχρηματοδότηση αγροτοπεριβαλλοντικών και κλιματικών καταβολών ε, και δι' στην βιολογική γεωργία. Η η μείωση, α, η, μείωση αυτή δεν θα πρέπει να σημειωθεί σε περιοχές όπου έχουμε αντιστασμιστικά μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Ε, εάν θέλουμε να αντιστασμίσουμε την κλιματική αλλαγή, παραδείγματο χάρη αυξάνοντα ε, τι χορτολιβαδικές εκτάσει, ε, δεν θα είμαστε επιτυχημένοι. Δεν, δεν συνδέονται άμεσα αυτά αυτά τα δύο μέτρα σε μια οικονομία ε, χαμηλών ε, εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακο πρέπει να εφαρμόσουμε πλέον μέτρα τα οποία θα έχουν και κοινωνικές επιπτώσεις. Παραδείγματο χάρη στην κατανάλωση. Πρέπει να βελτιώσουμε την οτροπία κατανάλωσης προς τις νέες πολιτικές. Πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε τα ίχνη της ε, ενεργειακής ε, κατανάλωσης, ε, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά και δει στο διοξίδιο του άνθρακα. Εγώ υποστηρίζω έντονα ότι περιβαλλοντικά μέτρα θα πρέπει να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό μέχρι, του, μέχρι ε, ε, το, το στο 25% έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περιφέρειες με οικολογικό δυναμικό. Και τα συμπεράσματά μου είναι τα εξής. Οι κίνδυνοι αυξάνονται οι αποφάσεις στο, στο Durban ε, για την ε, μείωση, για την περιορισμό των κλιματικών αλλαγών μέχρι του ύψους των 2 βαθμών Κελσίου μάλλον θα αποτύχουν και η σημερινή μεταρρύθμιση ε, της ΚΑΠ με τα προτινόμενα μέτρα δεν προσφέρει ακριβώς τις καλύτερες ευκαιρίες για μια ομαλή προσγείωση στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Φίλιος, ο κόσμος μας. Πρέπει να μετακινηθούμε από ε, την, ε, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στις συγκεκριμένε περιφέρειες σε μέτρα τα οποία στοχεύουν στην εξασφάλιση των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των πρώτων υλών. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους μετρήσιμους στόχους αγροτικούς για το 2020 αλλά και μετέπειτα. Τα μέτρα πρέπει να είναι να στοχεύουν σε ξεκάθαρους ε, στόχους, να, να ε, έχουν λοιπόν σαφείς στόχους ε, και να αναποσανατολίζονται σε μια συγκεκριμένη μελλοντική εικόνα της γεωργίας μετά το 2020. Πρέπει επίσης να μειώσουμε, να κάνουμε ένα phase out στις άμεσες πληρωμές και να ε, σεβαστούμε τις, ε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και να τις μετρήσουμε με μια δελεχή ανάλυση. Ευχαριστώ την κυρία Φρέν Πάουερ και τώρα δίνω το λόγο στον καθηγητή Μπάκουαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που με επιτρέπει να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Ήδη ακούστηκαν πολλά πράγματα και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την αηφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τις δυνατότητες που έχουμε να τις βελτιώσουμε. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τρεις εναλλακτικέ λύσεις, τρεις προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, διαβούλευση το 2010 με την κοινή γνώμη. Αν κατανομή στα πλαίσια της ΚΑΠ και νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητη αλλαγή. Θα πρέπει να γίνει διαφορετική κατανομή των ενισχύσεων για τη Γεωργία. Διότι δεν χρειάζεται να γίνει πλήρης αναδόμηση. Είναι απαραίτητο να γίνει ανακατανομή. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μια, ένα πρασίνισμα της ΚΑΠ. Και τελικά, τι θα πρέπει να γίνει για να πάει καλά η Γεωργία. Να μην δίδονται πλέον οι άμεσες ενισχύσεις. τρίτη πρόταση, τρίτη ε, εναλλακτική λύση είναι κάτι το οποίο τα περισσότερα κράτη απέρριψαν. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να επικρίνει την Κομισιό. Και η μοναδική της λύση ήταν να ακολουθήσει την δεύτερη. Είπαμε ότι έγιναν επικρίσεις διότι δεν ήταν η ε, φιλόδοξη πρότασή της. Τώρα εφόσον έχουμε αυτή την ε, πρόταση της ενοποίησης να τη βελτιώσουμε. Ανακατανομή λοιπόν, πρασίνισμα της ΚΑΠ και καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων, κυρίως εξετάζοντας πώς θα μπορέσουν να διαρθρωθούν οι δραστηριότητες οι γεωργικές, πώς θα μπορούσαν να μειωθούν οι καταβολές μεγάλων κονδυλίων και πώς θα μπορέσουν οι νέοι γεωργοί να βοηθηθούν. Κατά την άποψη όμως το κύριο θέμα είναι το πρασίνισμα. Και αν δεν κάνουμε κάτι το σημαντικό στον τομέα αυτό, θα έχουμε χάσει την δυνατότητα που μας προσφέρεται να επιτύχουμε μεταρρύθμιση. Ποιοι είναι οι στόχοι της ανάπτυξης υπαίθρου. Στόχος είναι να έχουμε καλύτερη βιοπικιλότητα, προστασία των υδάτων και του κλίμακτος, αλλά θα πρέπει να δούμε κυρίως ότι με τον περιορισμό των κονδυλίων κινδυνεύουν κάποιοι πυλώνες να παραγνωριστούν. Εάν ε, δαπανηθούν τα πάντα στα πλαίσια του προορισμού για τον πρώτο πυλώνα και εγκαταλειφθούν δεύτερο και ο τρίτο, θα είναι λαθασμένη η προσέγγιση μα. Πράγμα που σημαίνει ότι τελικά δεν θα πάρει περισσότερα κονδύλια από ό,τι σήμερα η Γεωργία. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με λιγότερα κονδύλια. Άρα θα πρέπει να έχουμε καλύτερες ιδέες για να υποφελήθουμε τα χρήματα. Γιατί θα πρέπει να πρασινίσει η ΚΑΠ, διότι πολλοί λένε ότι αρκετά πράσινη έχει γίνει. Η Γεωργία δεν χρειάζεται περισσότερο να πρασινίσει. Η Ανέτ μας μίλησε για κάποιες θεωρητικές περιπτώσεις που αφορούν την ΚΑΠ και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα πρέπει η χρήση γης να είναι τέτοια ώστε να μπορέσει να προληφθεί και η διάβρωση των εδαφών. Και πολλοί λέγουν ότι η διαχείριση των ε, αρρώσιμων ε, επιφανειών θα πρέπει να είναι καλύτερη, πιο υφόρος για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη γεωργία. Υπάρχει επίσης η προσέγγιση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων που αποδεικνύει ότι υπάρχουν πάρα πολλές μη εμπορικές υπηρεσίες που παρέχονται μόνον από τους ε, ε, αγρότες και από αυτούς που ασχολούνται με την προστασία των δασών. Και οι περισσότερες τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν είναι εμπορικές υπηρεσίες, διότι και έτσι δεν θα πρέπει να μας σοκάρει το ότι όλο και περισσότερο διαβρώνεται το κεφάλαιο οποίο διαθέτουμε. Δεν είναι βέβαιο ότι οι κυβερνητικές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, είναι σοβαροί στο θέμα αυτό και δεν είμαι πεπισμένος ότι οι κύριοι δικαιούχοι το έχουν λάβει το θέμα αυτό σοβαρά υπόψη και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πώς θα επαναλαμβάνω να πρασινίσουμε την ΚΑΠ. Τους τελευταίους 20, τα τελευταία 20 χρόνια μιλούμε για αυτό το θέμα. Από όσον ξέρω εγώ, θέλουμε να το κάνουμε αυτό μέσω του δεύτερου πυλώνα, ε, σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τι γίνεται σε ε, επίπεδο συμβατικό και εθελούσιο, σε πολυετήσια βάση, με χρηματοδότηση και με ε, σο αξιολόγησης είχαμε στο παρελθόν κάποιες περιοχές οι οποίες δικαιούνταν ε, επειδή είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά ε, τα απαραίτητα στοιχεία, αλλά ό,τι έγινε στα πλαίσια του πυλώνα 2 δεν ήταν απολύτως επιτυχές. Ελέγχεται ότι πρόκειται για κάτι το εντελώ γραφειοκρατικό και αργό και βεβαίως ε, αυτό ε, ε, έχει σήμερα να κάνει και με το θέμα της συγχρηματοδότησης, γιατί με την οικονομική κρίση πολλές χώρες δεν μπορούν στα πλαίσια αυτού του πυλώνα να συνεχίσουν να συμμετοχωρηθούν δράσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την στρατηγική. Ε, με, από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο θέλουμε να ισχύσουμε τον, τον πυλώνα 2. Σήμερα όμως είναι ε, διαφορετικά τα πράγματα και επειδή δεν θα μπορέσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών να δοθούν περισσότερα κονδύλια στον πυλώνα 2, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε τον πυλώνα 1 να τον κάνουμε πιο πράσινο. Πώς θα τον κάνουμε πιο πράσινο. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιε είναι οι πολιετής δράσεις και ποιε θα είναι οι πρακτικές οι οποίες θα εντοπιστούν και θα χρησιμοποιηθούν και θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους γεωργούς ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις βιώσιμες πρακτικές. Αυτή η προσέγγιση είναι ε, ετήσια, απλή και έχει σαφή προτερήματα για όλους και πρέπει θα είναι κοινή και δίνει την δυνατότητα ίσως να είναι απλή και να εφαρμόζεται, είναι βασική, να εφαρμόζεται από όλους. Τώρα, η διαχείριση ε, του περιβάλλοντος μπορεί να υπακούσει σε τέτοιου είδους ε, βασικές αρχές. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να προσαρμοστεί και στις μεθόδους και στις κλιματικές ιδιομορφίες κάποιας, κάθε περιοχής. Άρα σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να διαχειριστεί κανείς έτσι το σύστημα. Και το θέμα είναι, μπορούμε να κάνουμε πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα και να καταλήξουμε σε εφικτά αποτελέσματα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η μεταρρύθμιση έχει κάποιες δυνατότητες να το κάνει, αλλά θα το πρέπει να το κάνει σε μεγάλες, μετά από μεγάλες ριζοπαστικές αλλαγές. Αν δείτε ε, τι σημαίνει ε, πρασίνισμα στον πυλώνα 1, θα πιστεύουν ότι οι πληρωμές θα πρέπει να Πρασινίσου ποσοστό 30%. Θα σας πω κάποιοι ότι αυτό το πράγμα τους φαίνεται ότι είναι δύσκολο. Τι χριστουγεννιάτικο δώρο θα τους κάνετε, ενώ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οι πάντες να προσπαθήσουν να κάνουν. Δυνητικά όμως αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη δυνατή, διότι 30% ε, του ποσοστού αυτού ε, πληρωμές πράσιμες σημαίνει 12,5 δις πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, πενταπλασιασμό των δαπανών για τη γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι αν θέλουμε να αυξήσουμε τις πόρους για να τους πενταπλασιάσουμε για την, το πρασίνισμα, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και πολύ καλή βελτίωση της διαχείρισης του όλου. Βλέπετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι τα πρακτικά μέσα που θα ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την πολιτική και να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι και κάνουμε επικρίσεις μόνο. Υπάρχουν σίγουρα ε, δυσκολίες. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε τις μη βιώσιες μονοκατηγέργειες. Θα πρέπει να προλάβουμε τη διάβρωση του εδάσους του εδάφους, με συγχωρείτε, την ε, μείωση των οργανικών ε, ουσιών του εδάφους και την μείωση της ε, μόλυνσης. Να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μια δυναμική διαδικασία, να έχουμε εναλλαγή των εσοδιών και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τους αγρότες στο να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις και να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές ώστε να υπάρχει κέρδος για το περιβάλλον. Πρέπει να πω ότι στην ε, μελέτη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ντροπή το ότι δεν γίνεται προσπάθεια να εξηγήσει κανείς ε, ποσοτικά τα ωφέλη αυτών των προτάσεων ε, για το περιβάλλον. Δεύτερον, δεύτερο μέτρο. Θα πρέπει να δίδονται ενισχύσεις στους μικρούς ε, γεωργούς, ε, κυρίως ε, και να διατηρούνται τα, οι, οι αγροτικές χορτολιβαδικές περιοχές στις ανατολικές χώρες, όχι και να μην γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Πρόκειται για ε, μέτρα τα οποία θα πρέπει να είναι λογικά και να μπορέσουν ε, να δοθούν κοινά ε, χαρακτηριστικά σε όλους, ώστε να μπορέσουν όλοι να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές βασιζόμενοι στο γεγονός ότι πρέπει να προστατεύσουν με τον ίδιο τρόπο τη γεωργία, το έδαφος και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Θα πρέπει να δοθούν λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες διευκρινήσεις, διαφορετικά αυτό το οποίο κάνουμε είναι με την αβεβαιότητα να προκαλέσουμε αρνητικές επιπτώσεις αντιθετικές. Το κλειδί για μένα, για να επιτύχουν αυτά τα πράσινα μέτρα είναι μπορούμε να επιστρέψουμε ε, σε αυτά τα οποία λέγονταν καταρχάς ε, ώστε χωρίς να εγκαταλείψουμε εντελώς τον πυλώνα 2 να μπορέσουμε να λάβουμε τα πράσινα μέτρα ώστε να γίνονται οι βιοκαλλιέργειες υποχρεωτικές στον πυλώνα 1. Πολύ ωραία. Τότε οι αγρότες οι οποίοι πραγματικά λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα ε, πράσινης γεωργίας και για του βελίούς του περιβάλλοντος και του κλίματος να θεωρείται ότι κάνουν κάτι με αυτό το οποίο είναι υποχρεωτικό για να μπορέσουν να γίνουν σωστά τα πράγματα. Και βεβαίως αυτή η έλεγχη θα πρέπει να είναι υποχρεωτική ώστε οι αγρότες οι οποίες συμμετέχουν σε τέτοιους προγράμματα να υποφελούνται και αυτοί οι οποίοι δεν είναι ή να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε μέσα ή να τους υποχρεώσουμε να κάνουν υποχρεωτικό πρασίνισμα. Αυτός ε, είναι ένα από του ε, διαθροτικούς τρόπους να προχωρήσουμε για να βελτιώσουμε τις προτάσεις. Παρόλο που δεν έχω περισσότερο χρόνο, σαφώ χρειάζεται περισσότερη ώρα να τα συζητήσουμε, αλλά καταρχά μπορεί οι προτάσεις αυτές να, να αντικαταπτρίζουν ένα σημαντικό βήμα μπροστά για την εξέλιξη της ΚΑΠ. Και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάκουελ. Ώρα των ερωτήσεων. Ο κύριος Μποβέ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις δύο παρεμβάσεις. Δύο ερωτήσεις. Σε καμία από αυτές για θέματα περιβαλλοντικά δεν τέθηκε το θέμα της κτηνοτροφίας εκτός εδάφους. Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει να κάνει με το περιβάλλον είναι αυτό της ε, κτηνοτροφίας χείρων ή πουλερικών εκτός εδάφους όπως λέγεται και έτσι βλέπουμε ότι πολύ μεγάλες ε, ποσότητες μπορούν να παραχθούν με πάρα πολύ επιζήμιες ουσίες. Και έτσι αυτό το θέμα της γέντρωση των ζώων είναι ένα θέμα σημαντικό για τη μεταρρυθμιστικά. Πείτε με την απόψή σα. Δεύτερο θέμα, ακούγοντας παρεμβάσει σας για το πρασίνισμα, πιστεύω ότι υπάρχει κάτι το παράδοξο που είναι πρόβλημα εδώ. Σήμερα ο πρώτος πυλώνας θεωρείται ως για τους γεωργούς ο πυλώνας ενίσχυσης του εισόδηματός τους το πρόβλημα της ε, ε, αποδοτικότητας δεν θα ήταν πιο ε, θετικό εάν οι γεωργοί παρήγαγαν και είχαν αυτό το σύστημα. Δηλαδή, είναι το σύστημα αρνητικό. Πρώτα οι γεωργοί ε, λαμβάνουν υπόψη την ενίσχυση για να αυξήσει το εισόδημά του και μετά παράγουν. Όσο είμαστε λοιπόν σε αυτό το μοντέλο, ποτέ δεν θα έχουμε πρασίνισμα αποτελεσματικό. Μήπως θα πρέπει λοιπόν, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αναφέρατε και στην προηγούμενη συζήτηση τώρα, μήπως θα πρέπει το εισόδημα να έχει σχέση και με τα ποσότητα των προϊόντων που πολλούνται και να αποδεσμευτεί όλο αυτό το θέμα που μιλούμε και αφορά το εισόδημα από το θέμα της καταβολής των ενισχύσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάιον. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις οι οποίες και οι δύο είχαν στόχο να, να αντιμετωπίσουν την ανάγκη μιας πιο πράσινης πολιτικής ε, σε συνδυασμό με την επίτευξη των στόχων της αηφόρου γεωργίας. Για να ε, επανέλθω τώρα στην πρώτη ομιλία η οποία ήταν εξαιρετική. Πιστεύω ότι το θέμα της αηφορίας και το να ληφθεί υπόψη σοβαρά στον πρώτο πυλώνα μπορεί να απαντηθεί ως εξής ο, ο προϋπολογισμός για τα τρόφιμα ε, και για την αγροτική παραγωγή πρέπει να αντισμετωπιστεί πολύ σοβαρά και για την ασφάλεια των ε, πρώτων υλών. Ε, εγώ προέρχομαι από τη Σκωτία και γνωρίζω αρκετά για την εκτινοτροφία αλλά και για την αγροτική παραγωγή θα πρέπει ο προϋπολογισμός για την κάλυψη της γεωργίας με επωφελείς ουσίες και χημικά στοιχεία να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αυτό αφορά κυρίως ας πούμε, λιπάσματα και περιεχόμενα ζωτούχων ουσιών. Ε, ευχαριστώ. Thank you very much. Um, my questions... Ευχαριστώ. Ε, εγώ απευθύνω την ερώτησή μου στην πρώτη ομιλήτρια η οποία με τρόμαξε. Και θα εξηγήσω γιατί. Λέτε ότι εμείς ως παραγωγή μπορούμε να επηρεάσουμε το κλίμα με πολιτικές αλλαγές που μπορούν και πολιτικές αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν μέσα σε αυτό το σώμα. Το κλίμα έχει αλλάξει και πέρσι το, το, ο καιρός στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τόσο κρύος, τόσο απέσιο ήταν το κρύο που κατέστρεψε τα δύο τρίτα της παραγωγής του, των τεφτλών. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις αυτών των πολύ κρύων και άγριων χειμώνων. Ε, το άλλο στοιχείο που, για το οποίο μιλήσαμε, για το άζωτο, είπατε ότι 10-20% των αζωτούχων ουσιών που ε, χρησιμοποιούνται χάνονται. Ε, εγώ διαφωνώ ριζικά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και αζωτούχων ουσιών. Εάν μειώσουμε κατά 20% θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγή ε, τον, την αγροτική παραγωγή. Διαφωνώ λοιπόν με την πρότασή σας για μείωση. Ευχαριστώ. Θα, θα είμαι σύντομη. Όταν ο καθηγητής κύριος Μπάκουελ είπε ότι κινδυνεύουμε να ενθαρρύνουμε ε, κακές αγροτικές πολιτικές, θα ήθελα να ρωτήσω, ε, λέει η κυρία Μαγκίνες, ποια είναι αυτά τα επιζήμια μέτρα. Δεύτερον, νομίζετε ότι η βιολογική γεωργία πρέπει να έχει ε, εν λευκό εξουσιοδότηση ανάπτυξης και χρήσης. Συζητήσαμε την ιδέα να επιτρέψουμε ε, παραγωγούς να αναπτύξουν διάφορα πράσινα μέτρα ή νομίζετε μόνο βιολογική γεωργία είναι πράσινη και ο καθηγητής κύριος Μπάκουελ απευθύνουμε σε αυτό. Νομίζω ότι τα σχόλια που είπατε είναι πάρα πολύ σωστά. Ίσως θα μπορούσατε να μας τα αναπτύξετε λίγο περισσότερο. Εμείς έχουμε μεγάλες ελπίδες όσον αφορά τις προτάσεις της Κομισιόν ότι θα αποφύγουν την, μεγαλύτερη επιδείνωση της αγροτικής παραγωγής. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν αυξάνεται, ότι δεν έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και Ζητούμε όλο και περισσότερες θυσίες από την κοινωνία, από τους πολίτες μας, αλλά ε, δεν ε, ε, προβλέπουμε στον προϋπολογισμό την κάλυψη των αναγκών και ζητούμε όλο περισσότερες οικονομικές θυσίες. Ο κύριος Σιτζίνσκι, συμμερίζεστε και δύο την άποψή μου ότι στην πρόταση για τη μεταρρύθμιση γίνεται αναφορά στα εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπο στο κλιματολογικό πρόβλημα, στην βιοπικιλότητα, στις πεταλούδες, στα πουλάκια, αλλά δεν μιλάει κανείς για δύο σημαντικά θέματα, για τη γη και για το νερό. Πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη, μιλούμε συνέχεια για την ανταγωνιστικότητα που είναι προϋπόθεση για να είναι κανείς αποδοτικός και ξέρουμε ότι η ανταγωνιστικότητα σημαίνει αντατικοποίηση δηλαδή παραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ενώ όταν μιλούμε για παραγωγή ένα εκτάριο, μιλούμε για εισοδήματα. Υπάρχει κάτι που ονομάζεται ακόμη ευρωπαϊκό πρότυπο της Γεωργίας, διότι το πρασίνισμα σημαίνει ανταδικοποίηση. Και η καινοτομία στη Γεωργία προσεγγίζει περισσότερο την ε, εντατικοποίηση ή περισσότερο το πρασίνισμα. Προς τα πού πρέπει να στραφούμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στον κόσμο και για να ανταποκρινόμεθα στην ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων ειδών διατροφής που παράγονται. Ευχαριστώ κύριος Λέντσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα να πείσω την προσοχή σας στο γεγονός το εξής. Συζητώντα για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και για το 30% πρασίνισμα του πρώτου πυλώνα, Επίτροπος και οι εμπειρογνώμονες μας είπαν ότι οι γεωργοί δεν θα έπρεπε να φοβούνται, διότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόμη και σήμερα, έχουν μη καλλιεργήσιμες γέες, μάλλον μη καλλιεργημένες γέες, για τις οποίες θα μπορούσαν να ζητήσουν ε, ε, επιδόσεις. Επιδοτήσεις, συγγνώμη. Ο μηχανισμός θα βοηθήσει ή θα σημαίνει μεγάλη γραφειοκρατία και άχθος και για την κάθε δίκαιση κράτους και για τον κάθε αγρότη. Θα ήθελα να συζητηθεί αυτό το θέμα περαιτέρω, διότι Θέλουμε να θεσπίσουμε μία λύση την οποία θα επικρίνουν και οι ίδιοι οι αγρότες και όπως λέγουν και οι εμπειρογνώμονες, το σχέδιο αυτό δεν είναι και πολύ αποδοτικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Εκεί στο βάθος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να, να χαιρετήσω αυτή τη συζήτηση και τους ε, εξαιρετικά, τους, τις εξαιρετικές ομιλίες από τους καθηγητές και τους εμπειρογνώμονες. Θα έχω μια ερώτηση, αλλά δεν αναμένω την απάντησή σας. Πιστεύω ότι είναι λάθος η μονομερής προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής. Διότι στο μέλλον δεν θα χρειαστούμε μόνο αγροτική παραγωγή, αλλά η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να καλύπτει συγκεκριμένα προβλήματα. Επισητιστική επάρκεια, πρώτες ύλες και σωστή ορθολογική χρήση της ενέργειας. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις εν ώψη αυτών που συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου καινούριε πολιτικές εφαρμόζονται, νέες τεχνολογίες ε, υψηλότερων αποδόσεων σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, πώς θα λάβουμε υπόψη τώρα αυτά που συμβαίνουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Τρίτον, η ορθολογική χρήση των πόρων μπορούμε να επιτύχουμε μια καλύτερη χρήση των πόρων, μπορούμε να πετύχουμε μια άμβληση, μια αντιστάθμιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, έτσι ώστε να αντισταθμίσουμε με συγκεκριμένα μέτρα τη ζημιά από την αλλαγή του κλίματος. Μιλάμε συνέχεια για την αλλαγή του κλίματος, αλλά ε, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια μέτρα χρειάζονται, όχι μόνο για να περιορίσουμε το, τα αέρια του, του θερμοκηπίου, αλλά να φτιάξουμε προϊόντα τα οποία είναι ε, πιο, ε, αντιστέκονται περισσότερο στις αλλαγές, είναι πιο δυνατά και επίσης χρειαζόμαστε μέτρα για τη διαχείριση των προβλημάτων αυτών νερό, γη και αέρας. Χρειαζόμαστε διαχειριστικά προγράμματα για τη βέλτιστη χρήση αυτών των πρώτων υλών των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ε, μιλάμε βεβαίως για τη βιολογική παραγωγή των οργανικών λιπασμάτων, αλλά βλέπουμε όλο και περισσότερα λιπάσματα να χρησιμοποιούν φόσφορο ε, και άζωτο. Ε, τα οποία ξέρουμε τι επιπτώσεις έχουν στην γεωργία. Έχουμε δει τις ζημίες που, που έχουν ε, προέλθει από τις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει ε, να ακολουθήσουμε όπως και η Βραζιλία ορισμένες καινούργιες πολιτικές. Η Βραζιλία έχει δώσει το παράδειγμα σε πρωτοπορία και καινοτομίες. Δεν αναμένω απαντήσει σήμερα, αλλά εκτός από τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν τώρα για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, χρειαζόμαστε και άλλες δέσμες μέτρων. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν καλώς έχει προτείνει αυτά που έχει προτείνει για το άμεσο μέλλον. Ε, είμαι ικανοποιημένος με τους ε, πόρους, με τους χρηματοδοτικούς πόρους και τα μέτρα που προτείνει για την ανάπτυξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης αλλά μην ξεχνάμε και τον πιο πρόθεσμο ορίζοντα. Ευχαριστώ τον Υπουργό Γεωργίας και της Ρουμανίας για την ερώτησή του και τώρα θα δώσω το λόγο στους δύο παρεμβαίνοντες για να απαντήσουν. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Φρίμπαουερ, Φράιμπαουερ, για τη δέσμη αυτή των ε, ε, ερωτήσεων και θα προσπαθήσω να τις ομοδοποιήσω σε τρία μέρη. Καταρχάς, ο πρώτος πυλώνας. Ρόλος του είναι να δίνει λεφτά στους παραγωγούς χωρίς να βελτιώνει ε, τα αποτελέσματα ή την παραγωγή έχουμε ορισμένες ε, λανθασμένες εντυπώσεις, ε, ιδίως όταν ο παραγωγός ε, καλλιεργεί εδάφη τα οποία δεν είναι δικά του. Συνήθως το εισόδημά του προσαρμόζεται στις, στις, νίκη που πληρώνει για τα εδάφη αυτά είναι ανάλογα με τις πληρωμές που λαμβάνει. Και βλέπουμε ε, τέτοιες κινήσεις στη Γερμανία έτσι ώστε να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος αυτών των άμεσων πληρωμών δεν είναι ε, καλή λύση. Δεύτερον, η εντατικοποίηση. Actually, um, um, what, uh, what really production... Αυτό το οποίο πραγματικά συμφιλιώνει την παραγωγή και το περιβάλλον μπορεί να είναι η εντατικοποίηση. Αλλά αναφέρομαι εδώ στην μετακίνηση από την τεχνολογία στη γνώση. Προς αυτό το οποίο αποκαλούμε οικολογική εντατικοποίηση. Χρειαζόμαστε μια ίδια ή μεγαλύτερη παραγωγή με λιγότερους πόρους, με λιγότερα μέσα και επίσης χρειαζόμαστε μία αύξηση του βαθμού αντοχής και ε, ε, ε, δύναμης, αν θέλετε, των προϊόντων με λιγότερη χρήση πρωτοπαραγωγικών πηγών. 10 με 25% των ευρωπαϊκών εκπομπών, ρήπου δηλαδή στην ατμόσφαιρα, οφείλεται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Και τέλος, πού επικεντρώνεται το περιφερειακό μας ενδιαφέρον και πού υπάρχουν τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα, σε ποιες περιφέρειες. Αυτό πρέπει να τα προσέξουμε. Βεβαίως ε, υπάρχουν ορισμένες, ε, ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση του προϋπολογισμού ε, και των κονδυλίων που θα στοχεύουν συγκεκριμένα στην αύξηση ορισμένων διατροφικών ουσιών. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι ακόμη υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ούτως ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες χρήσης των θρεπτικών ουσιών, ιδίως εκείνων που περιέχονται σε κάποιο είδου οργανικά περιτώματα των ζώων που ακόμα δεν αξιοποιούνται ως λίπασμα. Και πολλές φορές αυτό το οποίο λέμε ως 75% ε, αναπόφευκτη απώλεια του αζωτούχου είναι πάρα πολύ ως ποσοστό ή στην διατροφική ή στην αλυσίδα. Και αν μπορέσουμε επομένω το φόσφορο, αυτές όλες τις ουσίες. Και όλα αυτά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε με πολύ μεγάλη ωφέλεια. Ευχαριστώ. Επόμενος, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω και εγώ τώρα σε κάποιες από τις τεθήσεις ερωτήσεις. Ε, ο κύριος Ζωζέ Μποβέ ερώτησε κατά πόσον θα ήταν πιο σωστό εάν οι παραγωγοί θα μπορούσαν να συνδέουν το εισόδημα σε το πόσο πολλούν. Θα ήταν υπέροχο να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και θα ήταν ακόμα πιο καλό εάν ε, οι καταναλωτές ήταν πρόθυμοι να προτιμήσουν τα, την προστασία του, του περιβάλλοντος και όχι μόνο το, το, το φαγητό γιατί ακριβώς όσον αφορά τα λοιπάσματα εδώ πέρα έχει γίνει διαφοροποίηση, έχει γίνει κατά τιμή της αγοράς και εκεί έχουν πιστεί καταναλωτές να, να προτιμήσουν τους τρόπους παραγωγής που ευνούν το περιβάλλον. Όμως το πρόβλημα είναι ότι αυτό αφορά για σχετικά μικρή μερίδα των όσων, των όσων δαπανούν οι καταναλωτές για το φαγητό. Φυσικά παρουσίαση, θέση σε εμπορία είναι σημαντικά και άρα το πρόβλημα παραμένει το οποίο είναι ότι το περιβάλλον είναι ε, μια ε, τεράστια αυτή τη στιγμή αποτυχία χτυπητή μεγάλη αποτυχία και άρα θα πρέπει να δούμε πώς ε, θα πρέπει τις σχετικές υπηρεσίες να τις ονομάσουμε δημόσια αγαθά Όμω ό,τι και να κάνουμε η αγορά ποτέ δεν θα δώσει την επιθυμητή τιμή και γι' αυτό και χρειαζόμαστε αυτή την παρέμβαση οι οποίε υπόκειται να υποστηριχθούν από το κράτο, Οπότε και κατά κάποιο τρόπο και η ΚΑΠΑ είναι τμήμα αυτή τη χρηματοδότηση και υποστήριξη ή θα υποστηρίξει ο ιδιωτικό τομέα μέσω κάποιων προγραμμάτων όπω ε, είπαν οι προλαλήσαντε για τα νερά, για την ε, κατακράτηση του άνθρακα τελικά να μετακυλιστεί κάποιο, κατά κάποιο τρόπο το κόστος στους καταναλωτές. Και αυτό είναι κοινό προγραμματής εις όλα όσα ε, ακούσαμε απόψε, ότι δηλαδή θα πρέπει η ΚΑΠ να υποστηρίξει όλο αυτές τις είδους τις υπηρεσίες. Η ΚΑΠ γιατί η αγορά δεν θα το κάνει. Επίσης η κυρία Μαγκίνες μας ρώτησε για τις επιβλαβείς υπηρεσίες. Ε, όχι, δεν θέλεις να σου πω τα όσα βλαπτικά γίνονται, γιατί έχουν γίνει σε κάποιους δείκτες, σε κάποιες μεταβλητές, κάποιες βελτιώσεις, αλλά γενικά έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Διαάβρωση, ε, βλαπτικά ε, αέρια και υδατικές εκπομπές, οπότε και γι' αυτό και δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, δεν έχει νόημα το να διαφωνούμε σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τους στόχους και για αυτού του είδους ε, της επιβλαβείς υπηρεσίες. Το θέμα είναι πώς οι γεωργοί θα έχουν ε, την κατάλληλη αμοιβή, ούτως ώστε να μπορούν να πετύχουν όλα αυτά τα οποία επιθυμούμε. Τι θα γίνει τώρα με τη βιολογική γεωργία, βεβαίως ε, θα πρέπει να βοηθηθεί, όχι μην θέτουμε φραγμούς, ε, άνοιξε η πόρτα σε σχέση με αυτή την πρόταση όσον αφορά τη βιολική γεωργία. Άρα αυτή η λογική να, να, να πάει μέχρι το τέλος και να ακολουθήσουμε και όσους ε, όσοι επίσης ε, με την πρακτική τους ωφελούν το περιβάλλον και δεν ζητάνε και παραπάνω. Επομένως αυτό είναι μια πιθανή απλούστευση της πρότασης. Και επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό στο να πληρώνει κανείς κάποιους για να συνεχίζουν μια αγαθή ωφέλιμη πρακτική. Το πρόβλημα είναι όλοι οι άλλοι οι οποίοι δεν ακολουθούν αυτό το παράδειγμα και οι οποίοι και αυτοί απαιτούν όμως αντίστοιχες αντισταθμίσεις. Και επομένως ε, εδώ ήταν το πρόβλημα του, οι θέση του, του, Ηνωμένου Βασιλείου για αυτή τη μεταρρύθμιση. Και αυτό έχει σχέση και με το δημοσιονομικό πρόβλημα. Γιατί αν δεχτεί το επιχείρημά μου ότι το βασικό θέμα σε αυτή τη μεταρρύθμιση είναι το πρασίνισμα και αν προκύψει ότι όλες οι φρονικέ οργανώσεις, κυβερνητικές και μη μέσα σε αυτή την ιστορία λένε ότι όλα αυτά είναι βλακίε, όλα αυτά είναι περιεχομένου, τότε δεν κάνουμε τίποτα που να ωφελεί και έχουμε μία ΚΑΠ η οποία λέει ότι έχουμε 12 δις που ωφελούν το περιβάλλον, αλλά όμως αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα έχουμε περισσότερη υποτίμηση, περισσότερη αμάβρωση και επομένω θα έχουμε το αντίθετο το επιδικομένου. Επομένω, όλα αυτά σχετίζονται και με τα όσα έχουν λεφθεί για τον προπολογισμό. Ε, ούτε ωφελεί το να λέμε ότι δεν είναι επαρκή ο προπολογισμό, δεν θα πάρουμε ούτε φράγκο παραπάνω και ακούσαμε τι σημερινέ εισηγήσεις ότι ε, έτσι έχουμε ε, την ασάφεια όσον αφορά το 70% και αυτό είναι στην καλύτερη περίπτωση διπλωματικό για το θέμα είναι ότι έχουμε συμπίεση των τιμών αρχή του 90 και, και τώρα και πιο μετά μετά το 2000 οπότε τρέχουν έχουν είναι πολλοί οι τιμές οπότε αυτή τη στιγμή ε, δεν υπάρχει εδώ και πολύ και δεν υπάρχει η λογική των ε, αντισταθμίσεων και άρα χρειάζεται μια άλλη λογική. Και άρα η μόνη λογική που τώρα μπορεί να σταθεί είναι αυτή του δημοσίου αγαθού. Άρα αυτό είναι το μόνο ουσιαστικό που μπορεί να θεωρηθεί χειροπιαστό. Οπότε τώρα πάμε σε μία ερώτηση από κάποιον ε, Πολωνό ε, που ρώτησε αν θα πρέπει να διαβάσουμε ή να καθισχάσουμε τους γεωργούς ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο αυτό το οποίο του δούμε για το πρασίνισμα γιατί ε, πάνω κάτω τα ίδια κάνουν μέχρι σήμερα και από την άλλη μεριά είναι άλλοι που λένε ότι δεν πρόκειται να ε, ωφελήσει καθόλου αυτή η μεταρρύθμιση και ακριβώς αυτή είναι η λεπτή σοβία που πρέπει να τηρήσει η Κομισιόν. Τώρα, εν κατακλείδη, έχω να σας πω τα εξής, ότι το ζουμί από αυτήν την μεταρρύθμιση είναι έχουμε δώσει τώρα όθηση προς σωστή κατεύθυνση στην ΚΑΠ. Ακόμα αυτό, ακόμα αυτό δεν έχει κρυφθεί. Ε, το, πράσι, το πρασίνισμα ε, σωστό. Ε, το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα οποία σωστά επαγγελόμεθα, αν θα τα καταφέρουν πως πρέπει και βέβαια απόκειται και σε εσά το να μας βοηθήσετε και όλα αυτά να πάνε καλά. Bon, merci ο πρώτο, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάκλε. Και τώρα, η Καταρίνα ε, Σαζαβαλίνσκα, η Διευθύντρια του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη της Υπέθρου και την Ανάπτυξη της Ακαδημίας Επιστημών της Πολωνίας. Ε, θα λάβει το λόγο και κατόπιν ο Χεσούς Γκονθάλες Ρεχιδόρ από το Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσια της Μαδρίτης θα λάβουν τη σκητάλη σε σχέση με το βασικό θέμα της ε, ισόρροπης ε, ανάπτυξης της υπαίθρου. Thank you Καταρίνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έχουμε έτσι διαρθρώσει τα πάνελ, ούτως ώστε εγώ να σας μιλήσω κυρίως όσον αφορά τις βασικές θέσεις που, που, διέπουν την ανάπτυξη της υπέδρου σε σχέση με την διακυβέρνηση που είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Χεσούς περισσότερο θα σας πει όσον αφορά άλλες πτυχές. Oh, Οπότε, για να δούμε τώρα αυτές τις βασικές έννοιες. Τι θα πει η εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης υπαίθρου. Να δούμε επομένω τι, τι περιεχόμενο έχει αυτή η έννοια, μην το αφήνουμε ω και, και κενή, έννοια, κενέ λέξεις και να δούμε και ε, κατά πόσον λείπει, υπάρχει σήμερα ισορροπία στην υπαίθρο σήμερα στην Ευρώπη και να δούμε μετά πώς, τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά και κατόπιν ε, να δούμε αυτού του είδου ε, οι πολιτικέ πώ θα βελτιωθούν μια που τώρα έχουμε το θέμα της ισορροπίας. Τελευταίο τώρα, αλλά σημαντικό, πώς θα γίνει σχετική διακυβέρνηση, πώς θα εφαρμόσουμε ε, στην πράξη αυτές τις ε, αρχές επαγγελίες για την εξισορροπημένη ανάπτυξη. Οπότε, για να δούμε αυτή η εδαφική προσέγγιση ε, προϋποθέτει ότι σημείο αναφοράς είναι ο τόπος, η τοποθεσία και όχι ο κλάδος, ο τομέας. Επομένω, το ένα είναι ευρωπαϊκή, το άλλο είναι αμερικανική προσέγγιση. Επομένως ε, το να μην λαμβάνεται υπόψη η τοποθεσία σημαίνει ότι κάνει κάποιο κάποια δουλειά και μετά πάει αλλού. Οπότε και η σχετική πολιτική υποστηρίζει του πιο πολλά υποσχόμενου κλάδου. Εδώ στην Ευρωπή έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή ότι η πολιτική αφορά ε, κάποιου τόπου όπου ήδη λαμβάνει χώρα και αυτού και στηρίζει, άρα είναι τελείω διαφορετική η προσέγγιση αυτή από την Αμερικανική. Επομένως, είναι πάρα πολύ βασική και αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πάνε παραπέρα από τη, τη, διοικητική αντιμετώπιση και αυτό γίνεται. Εδώ πέρα υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση και ο, δεν υπάρχουν επομένως γραφειοκρατικά διοικητικά όρια, περιορισμοί. Επομένως αυτό σημαίνει ότι οι τοπικά εμπλεκόμενοι ε, ε, συμμετέχουν και έχουμε αποκέντρωση τέλο πάντων από τη βάση προς τα πάνω, συμμετέχουν όλοι και οι τοπικοί θεσμοί, οι ντόπιοι είναι εταίροι, συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και, και έτσι θα πρέπει να κινητοποιείται η οι δυνατότητες ε, οι τοπικές και επομένως θα πρέπει έτσι να δούμε πώς θα έχουμε εξισορροπημένη πολιτική, και αγορές εργασίας, οπότε θα πρέπει να δούμε ε, ε, τι ανταγωνισμός υπάρχει για τις χρήσεις της γης. Το ανέφερε κάποιος συνάδελφος πριν, ότι ε, κοντράρει, δηλαδή ανταγωνίζεται η γεωργία με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οπότε άλλοι θέλουν να χρησιμοποιηθεί για οίκηση ή για ψυχαγωγία. Άρα η πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου βεβαίω και μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση του, της πολιτικής αυτής. Γι' αυτό λέμε για πολιτική που κάνει την προσέγγιση ανάλογα με την τοποθεσία και εξισορροπεί τα διαφορετικά στοιχεία. Για να δούμε όμως σήμερα τι έλλειψη ισορροπίας έχουμε είναι βασικό όπως λέει εδώ, όπως φαίνεται μάλλον εδώ αριστερά ε, ε, δεξιά και αριστερά το τι επιδόσεις έχουμε από τις διάφορες περιοχές της υπαίθρου στην Ευρώπη σήμερα και έχουμε εδώ τους εξής δείκτες που είναι τα όρια μεταξύ των καλών και των κακών μαθητών ε, πρόκειται επομένω πρώτα πρώτα για το θέμα της εξάρτησης από κάποιο κλάδο ή κάποιο τομέα μέχρι σήμερα επομένως έχουμε κάποιες περιοχές που εξαρτώνται τελείως από τη γεωργία και άλλους που ε, λιγότερο εξαρτώνται. Άρα εκεί που υπάρχει περισσότερη διαφοροποίηση από κάποιους τομείς όπως τον ε, δευτερογενή ή της υπηρεσίας ή κάπου να υπάρχει μείγμα των δύο ε, εκεί ακόμη τα πάνε πάρα πολύ καλά. Επίσης η δεύτερη διαχωριστική γραμμή που διακρίνει τους καλούς μαθητές από τους χειρότερους όσον αφορά τις περιοχές της ε, Υπέδρου είναι, Υπέδρου είναι η προσέγγιση, η εγκύτητα ή στις πόλεις. Οπότε υπάρχει ακόμα αυτή η μεγάλη διαφορά για αυτές τις περιοχές της Υπέδρου όπου δηλαδή είμαστε πιο κοντά στις ε, πόλεις θα πάνε καλύτερα από αυτές που είναι πιο περιφερειακές και για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι Αντιστοιχώς τώρα δεν έχω ένα χάραγα κάτι να σας ε, δείξω στο χάρτη, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι διαφορές, διαπιστώνουμε ότι ακόμα η Ανατολική Ευρώπη δεν τα πάει τόσο καλά στην Ήπεθρο από ότι η Μεσευρώπη ή η Δυτική Ευρώπη. Για να δούμε τώρα τις κάποιες νέες προτάσεις όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Θα αλλάξει, θεωρώ, δύσκολα αυτή η εικόνα μέσα χρόνια, ε, γιατί αυτές οι διαφορές είναι βαθιά ριζωμένες. Και, από όσο φαίνεται, οι κυβερνώντες δεν έχουν αντιμετωπίσει σωστά το πρόβλημα, γιατί εδώ, όπως βλέπετε, Έχουμε κάποιες περιοχές που τα πάνε ακόμα καλύτερα και δεν εξοντώς πολύ από τη γεωργία, αλλά ο δεύτερος πυλώνας κυρίως ασχολείται με τη γεωργία. Δεύτερον, Πρόκειται ακριβώς για την εγκύτητα προς τις πόλεις και εδώ έχουμε το, το αποτέλεσμα το οποίο μετακυλίεται από τη μία περιοχή στην άλλη. Δεν είναι θέμα λοιπόν εδώ πέρα αστικών κέντρων, αλλά ακόμα οι τοπικές και περιφερειακέ αρχές δεν έχουν αντιμετωπίσει σωστά το πρόβλημα. Έχουμε αυτή τη νέα πρόταση. Εδώ υπάρχει το μήνυμα ότι η, η πολιτική για τη γη και για την υπεθρο πανε πάνε χέρι-χέρι. Όμως, τι απόψει υπάρχουν. Υπάρχει συνένεση Επομένως, η ατζέντα λέει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κάθε περιοχή τα ε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Γι' αυτό και λοιπόν λέγεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφοροποίηση που υπάρχουν των διαφορετικών περιοχών της υπαίθρου. Η έκθεση Μπάρκα τι είπε, ότι εάν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αστιφιλία, τότε αυτό θα αποβεί αρνητικό και το οποίο επίσης είναι συνεπές με την άποψη ότι από σημεία του πολιτική θα και η απασχόληση. Όμως, από πλευρά της έκθεσης για την συνοχή προκύπτουν άλλα πράγματα. Ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να εξαπλώνεται από τις πόλεις στις λιγότερο εμπτυγμένες ε, περιοχές και πολλές φορές και στην Ήπεθρο. Άρα εδώ πέρα έχουμε διαφορές. Σύγκρουση ούτως υπήρχε μεταξύ περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής ε, συνοχής. Οπότε για να δούμε πώς θα πετύχουμε την επιθυμητή ισορροπία. Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ενιαία απάντηση στο ερώτημα αυτό. Άρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το πόσο κεντροκατευθυνόμενη θα είναι η λύση, ε, πόσο αυστηρότερη, πιο σφιχτή θα είναι η διαχείριση. Γιατί δεν νομίζω ότι θα πρέπει τη διακυβέρνηση να έχουμε ως επίκεντρο ως κεντρικό κριτήριο. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα συντεριάξουμε τους διαφορετικούς στόχους πολιτικής με τα διαφορετικά μέσα άσκησης της πολιτικής. Γιατί το θέμα είναι ποιοι είναι οι στόχοι της ε, τοπικής ε, διοίκησης. όσα προωθεί την πρόταση ότι δεν είναι πιο αποτελεσματική λύση οι επιδοτήσεις. Όμως θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία και άρα τα προγράμματα για την της υπαίθρου που χρησιμοποιούν πειραματικά οικονομικά μέσα πολιτικής, Φερρυπίν, στήριξη, επιδότηση νέων γεωργών. Αυτό γίνεται με βάση παλιότερα μοντέλα. Και καταλήγει να είναι ένα φάπαξ ποσό κατά αποκοπή σαν στήριξη στο εισόδημα. Μπορεί βέβαια να γίνει και να σχέδει και κάποια πολιτική που βασίζεται στις επενδύσεις. Αυτό τι θα κάνουμε έχει άμεση σχέση βέβαια με το τι αποτέλεσμα θα αποδώσει. Τώρα, για να δούμε τώρα. Πώς γίνεται η μέτρηση, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Έχουμε εδώ πέρα του τους τρεις τη ε, ΚΑΠ και έχουμε και κάποιους ε, νέους δείκτε μέτρησης αποτελεσμάτων αξιολόγηση που θα πρέπει να θεσπιστούν. Οπότε έχουμε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνηση και διαφορετικά προβλήματα. Η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες θα πρέπει να προσεχθούν και επίσης ε, κοινό πλαίσιο για την άσκηση της στρατηγικής μας να μην θεωρηθεί ότι με τους διαχωρισμούς των διαφορετικών πολιτικών θα πετύχουμε τίποτα. Το αντίθετο, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, συνέργεια των διαφορετικών πολιτικών και όχι διαχωρισμός αρμοδιότητων τώρα, όσον αφορά το Συμβούλιο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αρχέ οι αρμόδιε για την ε, ανάπτυξη, την περιφερειακή, ε, να μην είναι ένα και μόνο Υπουργείο αλλά βέβαια το θέμα είναι να μην υπάρχει αντίφαση, να μην υπάρχουν συγκρούσεις αρμοδιοτήτων, αλλά να υπάρχει συνεργασία. Οπότε, και τα άριστα των μέτρων με τους καλύτερους στόχους, με τα καλύτερα οικονομικά μέσα, εάν δεν εφαρμοστούν σωστά, δεν θα πετύχουν. Άρα, τότε συμπεράσματα. Από ό,τι φαίνεται, αυτού του είδους η στροφή προς την προσέγγιση με βάση κάποια τοποθεσία είναι το πιο σωστό. Κατά τη γνώμη μας, έχουν περισσότερες πιθανότητες έτσι, να άρουμε τις ανισορροπίες. Μόνο όμως όταν επιλεγούν τα ορθά μέσα. Εντοπίζονται οι ανισορροπίες και αντιμετωπίζονται και επιλύονται με, άειρονται με σωστά μέτρα. Και έτσι θα εκμεταλλευτούμε τις εγγενείς αλλά αυτό θα γίνει με συνεργασία, με συνέργεια και όχι με διάκριση αρμοδιοτήτων και διαχωρισμού. Βεβαίω και οι επιλέξιμοι θα χαρούν εάν δουν ότι υπάρχει τέτοιου είδου ε, συνέργεια μεταξύ ανάπτυξη και συνοχή, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών μέσων πολιτική των διαφορετικών ε, ε, των, ενισχύσεων, των επενδύσεων Και βέβαια θα πρέπει και οι γεωργοί να μπορούν να εμπλακούν όσον αφορά το τι θα γίνει με τον δεύτερο πυλόν και σωστή επίση επιλογή των αρμοδιοτήτων και περισσότερο να εστιάσουν την προσοχή μας στο αποτέλεσμα της πολιτικής, την εποπτεία, την αξιολόγηση και να μην προσπαθούμε να έχουμε περισσότερες δεσμευτικές, αυστηρές διοικητικές ε, διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων. αξιολόγηση που είναι το κλειδί και οι διαδικασίες που ισχύουν να είναι σε επίπεδο χώρας, σε εθνικό επίπεδο. Γιατί υπάρχουν διαφοροποίησεις μεταξύ διαφορετικών χωρών. Διαφέρουν δηλαδή, διαφέρει η διοικητική δομή των θεσμών οργάνων κάθε χώρας. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριος Γονθάλεφ. Eh, ευχαριστώ. Χαίρετε. Θα σας παρουσιάσω το PowerPoint αγγλικά. Αλλά θα σας μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για να είμαι σίγουρος ότι θα μεταφέρω πολύ σωστά τις ιδέες μου. Είναι ίσως αργά για σας κάπως, αλλά θα ήθελα στη σημερινή συζήτηση να παρουσιάσω μια κάπως διαφορετική πρόπτικη ή λιγότερο συμβατική από αυτή την οποία χρησιμοποίησαμε ως τώρα. Το πρόβλημα που πρέπει να τεθεί αυτή τη στιγμή είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις στην Ήπεθρο, σε κάθε περιοχή της Ευρώπης η ΚΑΠ. Ευνοείται η ισορροπία της Υπέθρου έτσι όπως εφαρμόζεται σήμερα η ΚΑΠ. Και δεν πρέπει να κάνει κάποιες προσαρμογές ώστε να με εξομαλυνθούν κάποιες ανισορροπίες. ανισορροπίες. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να παρουσιάσω την εξή ιδέα. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στην Ήπεθρο, στην Ευρώπη. Προφανώς σήμερα το απόγευμα μιλούμε τομεακά για το πρόβλημα. Έχουμε όμως ένα γενικότερο πρόβλημα με την ε, Ήπεθρο στην Ευρώπη και προσπαθεί να εισαγάγει η Επιτροπή μια νέα τεχνολογία για να διορθώσει την κατάσταση, πράγμα που επηρεάζει και ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που ζει στην Ήπεθρο. Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι το εξή. Παντού, σε όλες τις υπαίθριες περιοχές των διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση κάποιες ειδικέ περιοχές που έχουν παραδοσιακά μεγάλο γεωργικό βάσο, βάρος, το σχετικό οικονομικό βάζος της γεωργίας μειώνεται. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, διότι κάθε φορά που φτάνουμε σε υπαίθριες περιοχές και θέλουμε να τις μελετήσουμε, να τις γνωρίσουμε καλύτερα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μείωση της σχετικής οικονομικής δύναμης της Γεωργίας αρκετά σημαντική, πολύ σημαντική μάλιστα. Και αυτή η απώλεια συνοδεύεται δεδομένου τις περισσότερες ζώνες, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε μια γεωγραφική θέση στην οποία φαίνεται ότι η περιοχή όλη καλύπτεται από δραστηριότητες κτηνοτροφίας, ε, ε, δασών και γεωργία, βλέπουμε να υπάρχει μια κάποια ε, ουτοπία στις περιοχές. Διότι βλέπουμε ότι τα εισοδήματα προέρχονται από ποικίλε πηγές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Κάθε φορά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις περιοχές ζουν από εισοδήματα που τους αποφέρουν άλλες δραστηριότητες και όχι αμυγός η γεωργία ή η κτηνοτροφία. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο πρέπει να τεθεί είναι το εξή. Εάν η ΚΑΠ, ε, η, η, ΚΑΠ μάλλον ενισχύει ή όχι αυτές τις περιοχές όταν βλέπουμε ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στα πλαίσια της ΚΑΠ είναι εδαφικά αν θέλετε και γεωγραφικά πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Παραδοσιακά έτσι ήταν τα πράγματα. Παραδοσιακά λοιπόν η ΚΑΠ συγκέντρωνε τις προσπάθειες που κατέβελε σε κάποιες περιοχές. Λογικά στις πιο παραγωγικές, στα πλαίσια της ιστορικής εξέλιξης της ΚΑΠ. Άρα είναι πολύ συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα της ΚΑΠ ανάλογα με τις κάθε, την κάθε ζώνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει σχετικά μικρό αριθμό δικαιούχων. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξή. Παραδοσιακά η ΚΑΠ συνεισφέρει στην συνοχή ή όχι. Ενισχύει την έλλειψη συνοχής ή είναι πολιτική που οδηγεί στο να έχουμε πιο συνεκτικές περιοχές. Για να το αιτιολογήσω, θα σας πω μια φράση από τη δεύτερη έκθεση συνοχής. Τώρα είμαστε στην πέμπτη έκθεση. Στη δεύτερη, το 2001, ελέγεται το εξής, παραθέτω. Οι επιπτώσεις της ΚΑΠ είναι αρνητικές στις ζώνες τις πιο, ε, τις λιγότερο γόνιμες, τις πιο προβληματικές. Αυτό ελέγχθη και μελετήθηκε και οι εκθέσεις συνοχής, πρέπει να πω ότι από αυτού του θέματος επιδεινώθηκαν πάρα πολύ. Διότι έγινε μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση από αυτού του θέματος και κατέληξε το συμπέρασμα ότι μετά την μεταρρύθμιση του 2003 δείχνουν οι αναλύσεις ότι σε θέματα συνοχής τα πράγματα έγιναν πιο φτωχά κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε. Με αυτή τη γραφική παράσταση την οποία βλέπετε από την τελευταία έκθεση που αφορά τις υπαίθριες περιοχές και το έχετε σίγουρα δει, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να υπάρχει εδώ μία σύνθεση της που υπάρχει μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης κάποιων υπεθρίων περιοχών κάποιων χωρών σε σχέση με το μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Ανάλογα με, τον, ε, με τα κράτη που αναλύουμε, η απόσταση μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Οι πιο υπαίθριες περιοχές, αν θέλετε, οι πράσινες, κυρίως υπαίθριες, είναι 30% σε θέματα μέσου εισοδήματος κάτω από το μέσον όρο. Οι μέσες 10 ε, μείων και οι αστικές περιοχές 25 επάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ε, διαφορά μεταξύ των διαφορών ζωνών. Διότι έχουμε αρκετές ζώνες που είναι 30 με 40% κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Και εδώ μιλάμε για την ε, Ευρώπη των 27 και έχουμε να κάνουμε στατιστικές. Εάν μιλώ για χώρες πριν από την τελευταία ε, διεύρυνση, τα πράγματα αλλάζουν. Α δούμε τους παλιούς, τα παλιά ευρωπαϊκά κράτη, τα 15. Βλέπουμε μικρότερες αποκλήσεις. 91, ε, ενώ τώρα έχουμε 90 στο μέσο όρο. Και αν δούμε τι γινόταν στην ε, Ευρώπη των 12, έχουμε τρομερές αποκλήσεις. 60-50% αποκλήσεων. Τι σημαίνει αυτό, ότι πολλές ευρωπαϊκές υπαίθριες ζώνες βρίσκονται σε σχετική φτώχεια όσον αφορά τις ε, περιοχές της υπαίθρου που είναι κυρίως ε, γεωργικές περιοχές, διότι έχουμε αποκλήσεις του 40-50%. Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό λοιπόν ε, στην Ευρώπη με το θέμα αυτό ή δεν υπάρχει. Αυτό είναι το ερώτημα θέλετε. Και πώς βοηθάει η ΚΑΠ στο να αμβληνθεί αυτό το πρόβλημα. Η ΚΑΠ αυτή τη στιγμή, αυτή την οποία θέλουμε τώρα να μεταρρυθμίσουμε, απέκτησε σιγά σιγά αυτά τα προβλήματα. Εγώ βασίζομαι σε δύο επιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί έγιναν λάθη. Πρώτα απ' όλα διότι γενικά δεν ήταν τομεακός ο εστιασμός που θέλουμε να κάνουμε και δεν ελήφθη υπόψη το θέμα των ιδιαιτεριοτήτων κάθε περιοχής. Δεύτερον, βασικά, όσον αφορά την συμμετοχή της ΚΑΠ στην ανάπτυξη της υπαίθρου στα πλαίσια του δευτέρου πυλώνας όπως λέγουμε δεν μπόρεσε να καλύψει όλους τους δικαιούχους αλλά ένα τμήμα αυτών λίγους α, τους γεωργούς θα μου πείτε ότι υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση οι άξονες 3 και 4 αλλά βλέπετε τώρα σε μια άλλη γραφική παράσταση θα σας δείξω ότι αυτοί οι άξονες ήταν πραγματικά ε, Αμελητε. Το 3 δεν είχε οικονομικές ε, επιπτώσεις και δεύτερο, ο τέταρτος είχε μία ελάχιστη συνεισφορά στο δεύτερο ΛΟΝΑ. Άρα δεν έχουμε μεγάλο επηρεασμό τους. Και τελικά, ποιο είναι το συμπέρασμα. Η πολιτική για την ύπεθρο που έχουμε είναι ανεπαρκής σαφώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε αν δούμε την γραφική αυτή παράσταση που αφορά την ε, αναάξονες τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπετε τι συμβαίνει με αυτούς τους τρεις άξονες. Τώρα δεν θα πω σε λεπτομέρειες ανάλογα με τη χώρα, αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι χώρες τη δική μου, η Πορτογαλία ή τα νέα κράτη-μέλη, τον πρώτο άξονα στο δεύτερο πυλώνα, που ήταν ο πλειοψηφικός. Ο δεύτερος άξονας αυξήθηκε, ήταν δεύτερο σε αύξηση. Και εμένα αυτό το οποίο με απασχολεί είναι ο τρίτος, το μπλε. Το τρεις, οι άξονε 3 και 4, που παρέμειναν ε, μειοψηφικοί σε όλες τις χώρες, χωρίς καμία εξαίρεση. Πράγμα που σημαίνει ότι ο μέσος όρος για τα κράτη των 27 είναι 20% του δεύτερου πυλώνα, γι' αυτό το οποίο θα ονομάζαμε εμείς την πιο πολυτομεακή πολιτική. Το 20% του δεύτερου πυλώνα, κάνοντας με μικρό υπολογισμό, φτάνουμε στο 20% του 15%, δηλαδή μιλούμε για 2-3 εκατοστιαία ποσοστά όλου του προϋπολογισμού που δίνεται στην ΚΑΠ για μια πολυτομεακή και γεωγραφικά εδαφική ε, πολιτική της ΚΑΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ήταν ανεπαρκές το σύστημα που εφαρμόστηκε. Και λίγο προσέξαμε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Λίγο το προσέξαμε από αυτή την ε, οπτική γωνία. Η ΚΑΠ, λοιπόν, ήταν όλη η πολιτική της Ευρώπης για τη Γεωργία. Τώρα έχουμε τη νέα πρόταση. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την κατάσταση, τι προτείνει και τι λύσεις προτείνει η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι σημαντικά και όντως αποτελούν πρόοδο. Υπάρχουν ε, δύο-τρία σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε έξι νέες προτεραιότητες, ενώ στο παρελθόν είχαμε τέσσερις άξονες. Τα κράτη-μέλη μπορούν να συνάψουν μία συμφωνία για να αποφασίσουν και να καταγράψουν που εστιάζουν την προσοχή τους. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να λάβουν πρωτοβουλία τα κράτη-μέλη. Και τρίτο, και αυτό είναι το πιο καινοτόμο αν θέλετε, εμφανίζεται καλύτερο συντονισμός με τον πυλώνα 1 και κυρίως εμφανίζεται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί κανείς από όλους πόρους. Αυτή, αν θέλετε, είναι η μεγάλη καινοτομία. Μεγάλη και με την καινοτομία για σήμερα. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση που πήγαμε το 1999. Αλλά στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Το 1999 είχαμε μια πολιτική συνοχή από την οποία εξαρτόταν βασικά ε, για τρία από τα τέσσερα προγράμματα η ΚΑΠ. Έτσι λοιπόν σήμερα τι βλέπουμε κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις, παρά το γεγονό ότι εσφαλμένα λέγεται ότι είναι νέες προτάσεις. Και το ερώτημα είναι, τι σημαίνει συγκεκριμένα η συνεισφορά από άλλους πόρους. Διότι δεν βλέπουμε νέα μέτρα στα πλαίσια αυτού του νέου κανονισμού. Μιλούμε για συντονισμό μέτρων, μέτρων τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πυλώνα 2 και δεν είναι επαρκή. Άρα έχουμε να κάνουμε με μια μεσοβέζικη λύση. Είμαστε κάπως καλύτερα, αλλά όχι και πάρα πολύ καλύτερα. Κάτι άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον εδώ είναι το πρόγραμμα και η μέθοδος Leader. Πολλοί θα πούν ότι το έχουμε το Leader και το είχαμε και στο παρελθόν. 5% του προπολογισμού του δεύτερου πυλώνα πηγαίνει στο Leader. Όπως πολλοί που παρακολουθούν αυτό το πράγμα, πιστεύω και εγώ ότι οι δυναμικότητες και οι δυνατότητες του Λίντερ είναι πολύ περισσότερες από αυτές που του προσδίδουμε και από αυτό που θέλουμε να σώσουμε το 5%. Είναι πολύ πιο ε, σημαντική η συνεισφορά του Λίντερ εάν θέλουμε να την κάνουμε σημαντική. Και βεβαίω στο πλαίσιο αυτή τη μεταρρύθμιση υπάρχουν και αδύνατα στοιχεία τα οποία θα αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι και στην ίδια την έκθεση αξιολόγηση. Εάν γίνει προσεκτική αναθεώρηση του παραρτήματος 4 που αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, θα δείτε ότι υπάρχουν αμφιβολίες για τις επιπτώσεις αυτές. Ακόμη και η ορολογία που χρησιμοποιείται μπορεί να οδηγήσει σε ερωτηματικά. Υπάρχουν σαφείς προοπτικές μετά τη μεταρρύθμιση για την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου. Εγώ το διάβασα προσεκτικά το ότι λέγεται σε αυτό το παράρτημα. Και δεν βλέπω να είναι όλα πολύ θετικά. Αυτά τα ερωτηματικά μου δημιουργεί προσεκτική ανάγνωση αυτού του παραρτήματος. Διαρωτώμεστε λοιπόν, με αυτή τη μεταρρύθμιση θα προχωρήσουμε και όπως ελέγχθη στην αρχή θα βελτιώσουμε την συνοχή των υπευθείων περιοχών, αυτό το 90% που ελέγεται, ή θα συνεχίσει το θέμα αυτό να παραμένει άλυτο για το μέλλον. Διότι στην πραγματικότητα πολύ λίγα χρήματα παίζονται εδώ. Πολύ λίγα για το πρόβλημα που έχουμε και για το πώς είμαστε. 14 εκατομμύρια το χρόνο. 14 δις, με συγχωρείτε, είναι πολλά λεπτά, αλλά σε ε, σχετικούς αριθμούς, αλλά αν θέλετε όσον αφορά το θέμα το οποίο θέλουμε να λύσουμε σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτά αποφάσισαν, αυτοί πάνε τις αποφάσεις στην Ευρώπη. Από τις έξι λοιπόν προτεραιότητες που τίθονται εδώ, η έκτη μόνο ασχολείται με το θέμα αυτό εγώ δεν θέτω σε αμφισβήτηση την σημασία των άλλων προτάσεων. Είναι πολύ σημαντικέ. Απλώ υπογραμμίζω ότι αυτή η έκτη δεν έχει τύχει τη κατάλληλη μεταχείριση στα πλαίσια αυτή. Έτσι. Εκεί καταλήγω, σε αυτό το συμπέρασμα. Και τελειώνοντα, αναφέρω ότι έχουμε πρόβλημα. Διότι δεν έχουμε μια πραγματική ΚΑΠ και η πραγματικότητα είναι ότι λείπει μια τέτοια πολιτική και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε μια ισχυρή ΚΑΠ και δεν έχουμε μια ισχυρή πολιτική για τη γεωργία. Και κοινή πολιτική και πολιτική γενικότερα. Μία από τις δυνατότητες είναι το σενάριο της ολοκλήρωσης που αναφέρεται στην πρόταση αυτή. Το ερώτημα όμως είναι αυτός ο στόχος ενοποίησης για πότε προβλέπεται. Εφόσον ήδη έχουμε πει ότι το 1999 είχαμε ήδη μπροστά μας το σενάριο της μεγαλύτερης ολοκλήρωσης. Έλεγε κάποιος συνάδελφος, σιγά σιγά, στην Ευρώπη πάμε σιγά σιγά, το 2020. Το 2020 είναι πολύ ε, μακριά για τις σημερινές πρόπτικες. Κάνουμε λοιπόν μία ψευδοπολιτική ανάπτυξη της ε, υπαίθρου εδώ και κόσμου. 30 χρόνια ε, ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια πραγματική πολιτική ανάπτυξη της υπαιθρου εδω και κοσμου 30 χρονια ελπιζουμε οτι θα εχουμε μια πραγματικη πολιτικη αναπτυξη τη υπαιθρου Και ποια είναι η αμφιβολία μας. Αυτός ο μοναδικός, ο εγκάρσιος κανονισμός που αφορά τα ταμεία είναι η κατάλληλη απάντηση στα ερωτήματά μας. Ναι ή όχι. Είναι πολύ πολύπλοκος αυτός ο κανονισμός. Και θα δείτε ότι θέτει ε, προβλήματα και δυσκολίες διοικητικές τρομερές. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν αυτά που λέγονται. Λοιπόν, λίγα λεπτά, πολύπλοκος κανονισμός και μας απασχολεί αυτή η πολυπλοκότητα. Τελικά τι κάνουμε, ασχολούμαστε με ένα κανονισμό τόσο πολύπλοκο για να μοιράσουμε ψίχουλα σε κάθε περιοχή. Και το θέμα είναι πόσα λεφτά ζήνονται σε κάθε υπαίθρια περιοχή, σε κάθε ζώνη που θέλει να βελτιώσει την κατάστασή της πόσο θα πάρει η κάθε περιοχή και η κάθε ζώνη στο τέλος αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας. Και θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για περιφέρειες, για περιοχές όπως λένε οι στατιστικές. Για την ανάλυση ναι, αλλά για την ε, εφαρμογή, για το implementation δεν μπορούμε απλώς να μιλούμε για περιοχές όπως το NATS 3 Φερρυπίν, όπως το ονομάζουμε. Χρειαζόμαστε το επίπεδο ΝΑΤΣ 4 τουλάχιστον ζώνες και υπαίθριες περιοχές σε επίπεδο ε, διαμερισμάτων, υποδιαμερισμάτων με ομοιογενή στοιχεία. Όχι όπως τα πλαίσια του Λίντερ ζώνες που έγιναν με τεχνητό τρόπο και είναι ετερογενείς και δεν είναι αποδοτικές. Και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν για την ανάλυση. Ε, την ανάλυση μας βοηθάει η έκθεση, αλλά όχι για την εφαρμογή στην πράξη. Αλλά μια τέτοια ανάλυση είναι χρήσιμη, διότι βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλομορφία. Έχουμε ένα μοζαϊκό διαφορετικών ζωνών. Και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια ενιαία πολιτική αν δεν λάβουμε υπόψη ιδιαιτερότητες του κανενός. Και όταν έχουμε πολιτική η οποία βασίζεται σε τόσες αυστηρούς κανόνες, θα πρέπει να έχουμε ζώνες προς διαχείριση, οι οποίες να είναι ομοιογενείς μεταξύ τους, ενώ είναι ετερογενείς. Και τελειώνοντας, κάνω μια κάποια πρόταση ανάλυσης για να κάνουμε περαιτέρω. Τι χρειαζόμαστε. Μια ε, πολιτική υπερκανονιστική τύπου πρώτου πυλώνα, ένα πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή πολιτική για την Ήπεθρο. Ναι, πιστεύω. Βασικές προσανατολισμούς για την συγχρηματοδότηση εθνικών πολιτικών με τον κατάλληλο τρόπο και με, ε, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτερότητες του καθενός. Αυτό θέλω να προτείνω, διότι με αυτόν τον τρόπο αντιποκρινόμεθα στην πραγματικότητα. Ακούστε, τα περισσότερα κράτη-μέλη πριν από τη διεύρυνση έχει το καθένα τη δική του πολιτική για την υπεθρό. Και είναι πιο σημαντικό σε πολλές περιπτώσεις, εάν γίνεται αυτό που κάνει σε εθνικό επίπεδο, παρά αυτά τα οποία τους έρχονται από την Ευρώπη, όσον αφορά μέτρα και πόρους. Κοιτάξτε τους Άγγλους, τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τις κάτω χώρες, την Ιρλανδία, τα σκανδιναβικά κράτη, πρόσφατα την Ισπανία. Έχουμε εθνική πολιτική την ανάπτυξη της Πέθρου. Τι λείπει. Προφανώς η διαφοροποίηση, πρέπει να γίνει και ο διαχωρισμός μεταξύ της πολιτικής, της αγροεπισητιστικής και της προστασίας του περιβάλλοντος και άλλο είναι μια πολιτική εγκάρσια, πολυτομεακή που αφορά όλο το επίπεδο και αποτελεί ένα πλαίσιο γενικό με στο οποίο θα κινηθούν οι ε, πολιτικές κατευθύνσεις και αποφάσεις. Αυτό λοιπόν το οποίο τίθεται είναι η έλλειψη γενικότερου πλαισίου που δεν έχουμε, πώς θα δημιουργηθεί, Δηλαδή, ένα πλαίσιο γενικών προσανατολισμών χωρίς να τίθενται να αμφιβόλο οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και η πολιτική που θα κάνει κάθε χώρα. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε. Το μελέτησε το 2006 όσα και το ονόμασε νέο παράδειγμα ανάπτυξης της υπαίθρου και πιο πρόσφατα συμπληρώθηκε και από το... την πτυχή της αηφορίας. Και τι χρειαζόμαστε εν κατακλείδη. Κάτι το οποίο θα απλοποιήσει τους κανονισμούς ώστε η ΚΑΠ και η πολιτική συνοχής να είναι αποτελεσματικές για τις υπαίθριες περιοχές και την ανάπτυξη της υπαίθρου και τα εθνικά μέτρα που κάθε κράτο μέλος χρησιμοποιεί διαφορετικά να μπορέσει να εφαρμοστεί. Αυτή η εγκάρσια πολιτική που ονομάζω Rural Act θα πρέπει να αποτελέσει ένα πλαίσιο που χρειαζόμαστε όλοι. Και αν είχαμε και περισσότερους πόρους, τόσο καλύτερο. Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με θέμα πόρων, αλλά και με θέμα τάξης, με θέμα δόμησης των μέτρων που θα αποτελέσουν το γενικότερο λισάρι. Αυτά. Αυτό επομένως... Eh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τώρα ένα προβληματάκι. Ότι ο κύριος Υπουργός πρέπει να προλάβει μία πτήση οπότε να συνεχίσουμε έτσι με αυτόν μετά έχουμε ερωταποκρίσεις προς τους προσκεκλημένους μας και κατόπιν ε, ο Επίτροπος πρόκειται να δευτερολογήσει κλείνοντας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς, σε ένα δεκάλεπτο πρέπει να έχω φύγει. Όμως πρέπει πρώτα όλα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση διότι αυτή η συζήτηση ε, αποτελεί ακριβώς άλλη μία από αυτή τη σειρά των ε, συναντήσεων και θα πρέπει να εξηγήσουμε ή στους καταναλωτάς αλλά και ή στους γεωργούς το τι εστί αυτή η μεταρρύθμιση. Ε, ο καθηγητής μας ερώτησε για το τι γίνεται όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα στην γεωργία και τι γίνεται όσον αφορά τη διεθνή σκηνή. Ναι, Έχουμε διαρθωτικά προβλήματα, γιατί προβλήματα δεν έχουμε αρκετή ανταγωνιστικότητα. Και υπάρχουν οι λόγοι που γέννησαν αυτά τα προβλήματα και είναι ακριβώ το σύστημα των αμέσων πληρωμών. Δυστυχώ, οι προτάσει για την αλλαγή των πραγμάτων ε, κρίνονται ανεπαρκείς, διότι ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε, διότι έχουμε πάρα πολλέ εκμεταλλεύσεις οι οποίες πλέον δεν προχωρούν ε, στον εξονισμό γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί όταν κάποιο παίρνει το 60% των αμέσων πληρωμών, γιατί, γιατί να ενδιαφέρεται ε, να κάνει κάποιο είδους ε, αλλαγέ. Μια που έχει τέτοιου είδους εισοδήματα. Τώρα αυτό το πρασίνισμα. Το πρασίνισμα στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα φέρνει ελέγχθη το περισσότερο πλέον μεσό και δεν είναι αλήθεια αυτό και έχουμε τώρα τους γεωργούς οι οποίοι δεν ε, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρασίνισμα και γι' αυτό και τελικά δεν θα υπάρχουν συμπληρωματικά τέτοιου είδου εισοδήματα. Απλώς θα υπάρχει παραπάνω προσπάθεια. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου και ρωτήσατε εάν έχουμε περισσότερες γέες που έχουν υποβαθμιστεί. Μην κολλάμε στο 75% των αμέσων πληρωμών που είναι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή, διότι το επίπεδο το οποίο αφορά τον δεύτερο πυλώνα, δεν μας οδηγεί σε καμία κατάτμιση των πόρων. Δεν υπάρχει αρνητική συνέπεια αυτές τις πληρωμές. Ναι, θα πρέπει να σας ενθαρρύνω όλους εσάς πάντως, οικονομολόγους, επιστήμονες, να αναλύσετε αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Να βοηθήσετε την ανάπτυξη των περιφερειών και των χωρών. Περιμένουμε πώς και πώς τις θετικές επικοδομητικές σας προτάσεις. Αυτές που θα οδηγήσουν σε μια ανταγωνιστική καινοτόμα πολιτική και όχι σε μια πολιτική που απλώς θα βασίζεται στην παραγωγικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε δύο συναδέλφους. Δύο συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν ερωταπαντήσεις. Ο κύριος Σεκίνης πρώτος. Obszary wiejskie charakteryzują się opóźnieniem w rozwoju. Stąd tak ważne jest Έχουμε και κάποιε περιφέρειε που υστερούν όσον αφορά την ανάπτυξη. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώ θα εναρμονίσουμε την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική ανάπτυξη τη υπαίθρου. Και αυτό ισχύει ε, το σούτο μάλλον, καθώς δεν έχουμε ε, απεριόριστους πόρους για την ε, πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου. Οπότε, φαντάζομαι να καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ συχνά το ερώτημα το οποίο να δίνεται το πόσο σημαντικός είναι ο δεύτερος πυλώνας για τις νέες χώρες μέλη. Εκεί υπάρχει σημαντική στέρηση. Τέλος. Θέλω κάτι άλλο να σας αναφέρω. Όλα αυτά τα οποία αναφέρονται δεν κάλυψαν το εξής. Κανείς δεν ανέφερε το θέμα τις εμπειρία που έχουν αποκομίσει από τα 50 χρόνια εφαρμογή της ΚΑΠ και το πώς αυτή η εμπειρία θα βοηθήσει για το μέλλον, για το 2020. Έχουμε τις λύσεις της ΣΠΑΚ, έχουμε αυτά τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην ε, ε γεωργική πολιτική, ακριβώς αυτά τα οποία θέλουμε να ενισχύσουν και για τις ε, χρηματαγορές και τις κεφαλαγορές, διότι έχουν εισδύσει και στο χώρο της γεωργίας οι κερδοσκόποι και αυτό έχει ως συνέπεια ένα σωρό αρνητικά για την ΚΑΠ. Επομένως, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό να λάβουμε υπόψη την διακήρυξη, δήλωση της Βαρσοβίας, της 6ης Δεκάτου 2011. Και γι' αυτό θεωρώ Νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικά είναι αυτά τα οποία ελέγχθησαν και γι' αυτό και θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Ας λάβουμε επομένω υπόψη και αυτή την διακήρυξη δήλωση της Βαρσοβίας. Ο κύριος Βίλκιν είχε οργανώσει τη συνάντηση, ο οποίος προέρχεται από το ίδιο πανεπιστήμιο όπως και η σημερινή μας πανεπιστήμια κυρία Ζαβανίσκα. Οπότε, σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή την απόλαυση την πνευματική που σήμερα μας προσφέρατε. Αυτά που είπατε είναι απολαυστικά, είναι απολαυστικά και πολλά θεωρητικής και πρακτικής. Οπότε, κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Sí, muchas gracias, señor por Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ομιλίες και επειδή έχουμε πρόβλημα χρόνου θα θέσω μόνο τέσσερα ερωτήματα. Καταρχάς, ο δεύτερος πυλώνας, παρόλα αυτά τα οποία είπατε, θα πρέπει να παραμείνει στη Γεωργία. Εμένω αυτό. Δεύτερον, πιστεύετε ότι θα πρέπει να προδιαγράψουμε με περισσότερη αυστηρότητα πόσα κονδύλια, πόσες πιστώσεις θα δοθούν στα κράτη-μέλη. Πιστεύετε ότι χρειάζονται πιο συγκεκριμένα επιθετικά μέτρα στο δεύτερο πυλώνα από πλευράς προϋπολογισμού. Τρίτον, συγχρηματοδότηση Εντάξει, ο πρώτος πυλώνας 100%, χρηματοδοτείται 100% από την Κομισιόν. Στο δεύτερο πυλώνα πιστεύετε ότι χρειάζεται συγχρηματοδότηση. Πρέπει να συμμετάσχουν και άλλοι. Υπάρχουν περιφέρειες στη Γερμανία που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο όλο σύστημα της συγχρηματοδότησης. Πρέπει να το συνεχίσουμε ή πρέπει να εξαρτάται η συγχρηματοδότηση από τους ε, στόχους. Και τέταρτον, οι περιφερειακές ε, οι περιφέρειες και ε, θα πρέπει να έχουν λόγο, θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία συναπόφαση, θα πρέπει να ακούγεται η φωνή των περιφερειών διότι δεν είναι δυνατόν η Κομισιόν να οργανώνει μέτρα ή προγράμματα για την στήριξη της υπέθρου χωρίς να ακούγεται η φωνή των περιφερειακών αρχών και των περιφερειακών παραγόντων. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αυτές οι περιφέρειες ε, πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε από τη μία πλευρά να προστατεύεται η δημοκρατία, από την άλλη πλευρά όμως να εμπίπτουν και στα μεγαλόπνοα προγράμματα της, της Ένωσης. Θα ήθελα να πω το εξή. Πρώτα απ' όλα είναι ανεξάντλητο το εγώ συζητητή στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβουλίου για την άρξη ΠΕΤ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμες για τις εξαιρετικές τους ε, παρουσιάσεις. Επιβεβαίωσαν και κάποια από τα δικά μας ερωτηματικά και τις απόψεις μας και μας είπαν ότι πραγματικά θα πρέπει το όλο θέμα να το μελετήσουμε κάπως πιο εκβαθέως και βεβαίω είναι ανάγκη να υπάρξει συμβαστική λύση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για να καταλήξουμε σε λύση. Υπάρχουν πολλέ αντιφατικά στοιχεία. Τα μέσα πάντα θα είναι ανέπαρκη. Οι αντιφάσεις είναι τεράστιες, αλλά υπάρχει ένα κοινό άξονα. Θέλουμε να φτιάξουμε μία πιο δίκαια ε, κάπου που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες των κοινωνιών μας και για μένα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση. Σας ευχαριστώ και σας λέω ότι είμαι στη διάθεσή σας εάν θέλετε να συμμετάσχω και εγώ στις συζητήσεις που θα γίνουν για την επίτευξη αυτής της συμβαστικής λύσης που τόσο επιθυμούμε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα εκ μέρους του ΕΛΚ να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, τους εξέχοντες εμπειρογνώμονες που μας παρουσίασαν όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις. Όμως ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό κύριο Σαββίτσκι, ο οποίος δυστυχώς έπρεπε να φύγει για την εξαιρετική του συνεργασία με την Επιτροπή Γεωργίας. Σας παρακαλώ να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου στον Υπουργό κύριο Σαββίτσκι. Ποτέ δεν είχα τη χαρά να συνεργαστώ τόσο επικοδομητικά με, τον με έναν άνθρωπο τόσο εμπειρογνώμενο όπως τον κύριο Σαββίτσκι και εύχομαι καλές γιορτές και καλή πρωτοχρονιά σε όλους που δεν είναι παρόντες και στους παρόντες. Ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Θέλω να σας πω ότι ε, ευχαριστώ που οργανώσατε αυτό το συμπόσιο, αυτή την εκδήλωση, διότι νομίζω ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους συζητητές. Εγώ δουλεύω σε αυτό το κέντρο της Αντισή Πέδρου και οπότε και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω 100% με το συμπέρασμα του καθηγητού Γκονθάλεθ ο οποίο τα παρουσίασε πάρα πολύ ωραία και ακριβώ ανέδειξε το ζήτημα τη ανάπτυξη Πέθρου και ότι αυτό θα, το πρόβλημα θα πρέπει να ενταχθεί, να συμφιλειωθεί στον προβληματισμό για την ΚΑΠ. Ε, μπορείτε τώρα να διαπιστώσετε το ότι έτσι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, τις με την Ήπεθρο ε, στα διάφορα κράτη-μέλη της ε, Ήπεθρου. Και γι' αυτό θα πρέπει μας κύριε καθηγητά θα ήταν δυνατόν να ε, μπορέσουμε να εκπονήσουμε μια πολιτική ανάδειξη της Ήπεθρου σε αυτό το πλαίσιο διότι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ε, μια τέτοια πολιτική. Μπορεί να τη συλλάβουμε μόνο ως εθνική πολιτική και ευχαριστώ και τον προτέρων για την απάντησή σα. Σα ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρο, κύριε κυρία Ζεβανίσκα και ο κύριος ε, Γονθάλης Αρχιδόρ θα δώσουν πάρα πολλέ τιμέ απαντήσει στι ερωτήσει που έγιναν. Και έχουμε τον κύριο Δεκάστο και τον κύριο Τσόλ. Θα τον λόγο. Ναι, ναι, ίσως βιάζεται να προλάβει το αεροπλάνο, οπότε... Δίνω το λόγο στον κύριο ρεγκιδόρ. Mm. ρεγκιδόρ. Πες το. Ναι. Κοιτάξτε. Ε, έχουν υποβληθεί δύο πάρα πολύ σημαντικέ ερωτήσει και άλλε και άλλε, αλλά οι πιο σημαντικέ είναι δύο. Δηλαδή, η πρώτη. Πώ θα έπρεπε να εντάξουμε την πολιτική ανάπτυξη τη υπαίθρου στα πλαίσια των κοινών πολιτικών. Πώς το πιο στο... Ε, ε, σας υπενθυμίζω ότι αυτή η προβληματική δεν είναι κάτι το καινούριο. Όσοι είμαστε κάπως ε, μεγάλοι, ήδη ε, τα έχουμε πει από το 2003, ήδη τα προβλήματα αυτά είχαν τεθεί τότε που είχαν δει τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ και τότε ε, είχε αναδειχθεί αυτή η λύση ε, και είχαμε πει ότι δεν είναι η πιο σωστή αλλά ήταν αυτή η λύση που είχε βρεθεί και γι' αυτό σας λέω ότι τότε ο κύριος Μπαρνία που ήταν ο τότε επίτροπος δεν είχε έρθει σε μια συνάντηση γιατί ε, μίλησαν τετάρτη και έφυγε και τότε και εγώ σκέφτηκα ότι αυτό είναι τέλος δεν πρόκειται να έχουμε κοινή πολιτική για την Ήπεθρο που να εντάσσεται στην ΚΑΠ. Ε, τώρα όμως η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι αυτή η λύση δεν ήταν πιο σωστή και ότι πέρασε αρκετό χρόνος και ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική θα πρέπει να δούμε τι έγινε μετά την διεύρυνση γιατί το πιο δύσκολο για όλους είναι οι πιο γεωργικές χώρες ε, αυτές που έφυγαν από την προηγούμενη φάση Μιλάμε για 80% είναι αφιερωμένο στην γεωργία, οπότε εωρείται αυτό το όριμα μια που βεβαίω αναμφίβολα σχετίζεται κάπου με την Ήπεθρο. Όμως αυτό το οποίο εδώ είναι το θέτημα είναι να έχουμε μια πολυτομιακή ε, ΚΑΠ που να, είναι, που, που, να μπορεί να καλύψει και θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από την σημερινή ιδέα πρόταση για τη μεταρρύθμιση. Κομισιόν, Κοινοβούλιο, όλοι θα πρέπει να δώσουν την απάντηση και να διαπιστώσουν ότι αυτά τα οποία σήμερα έχουμε δεδομένα δεν πρόκειται να αρκέσουν για το μέλλον. Δεν λέω ότι τα μέτρα αυτά είναι λάθος, όμως δεν αρκούν. Να, ποια είναι η σωστή απάντηση. Δεν νομίζω ότι ο εγκάρισιος κανονισμός, ο οριζόντιος κανονισμός θα είναι η λύση, διότι πρόκειται για κάτι πιο περίπλοκο από αυτά το οποίο είχαμε αντιμετωπίσουμε το 1999. Επομένως, σας απαντώ. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε καλύτερα τις εθνικές υπάρχουσες πολιτικές με ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ε, πιο σωστό όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική. Επίσης μια διευκρίνηση δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες ζώνες ΝΑΤΣ 4 αυτό το κάνει η Κομισιόν. Τα κράτη. Ξέρουν, ξέρουν τα κράτη καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα. Όμως, εάν οι βασικές καθυντήριες, τα μέτρα πλαίσιο, η συγχρηματοδότηση θα το κανονίσει γιατί φυσικά και τώρα πάμε για τη συγχρηματοδότηση σίγουρα. Οπότε το βασικό είναι η έκτη προτεραιότητα. Αυτή που τώρα έχει κάπως συρρυκνωθεί το 21, το 55, το 60 δεν έχουν ανέβηθει αρκετά αυτά δεν αποτελούν κοινή γεωρική ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι καλή, είναι πολιτική που επιδέχεται βελτιώσεις, ε, α πούμε για τα γεωργοδιατροφικά, αλλά αυτό δεν είναι κοινή γεωργική πολιτική. Θα σας τα λίγο γενικά, δηλαδή δεν έχουμε χρόνο για περισσότερες διευκρινήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο πρόεδρος και τελευταίο, ο σε όλου και ο ο πρόεδρος ο Δεκάστρο θα κλείσει. Ευχαριστώ. Δεν θα καταλήξω σε συναγωγή συμπεριστηματών από αυτή τη συνάντηση, γιατί πέρασε και ο χρόνος. Απλώς και μόνο θα πω το εξή. Σήμερα διαπιστώσαμε επίσης ότι μπροστά στην πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη, δεδομένου ότι μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τη γεωργία στην Ευρώπη, το θέμα της γεωργικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας της, της μόνης διαχείρισης των φυσικών πόρων συγχρόνως, που είναι η επιθυμία και η προσδοκία όλο και περισσότερων πολιτών και όλο και μεγαλύτερη προσδοκία, μας κάνει να πούμε ότι είναι σαφές ότι η ΚΑΠ είναι απαραίτητη, αλλά ίσως όχι επαρκής για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι προκλήσεις. Η φιλοδοξία μας και το καθήκον μας είναι να καταστήσουμε την πολιτική αυτή χρήσιμη ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Διαπιστώσαμε από τις διάφορες παρουσιάσεις επίσης ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στο χρήμα για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Ο προβληματισμός είναι σημαντικό στοιχείο αλλά όχι το μοναδικό για να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που τίθενται. Γι' αυτό θα πρέπει η καινοτομία και η έρευνα, η έρευνα, η βασική και η εφαρμοσμένη να συνεισφέρουν και η μεταφορά γνώσεων στους γεωργούς επίσης. Χρειαζόμαστε επίσης τα μέσα που θα επιτρέψουν σε όλους τους εμπλεκόμενους στην διατροφική αισθία να χρησιμοποιήσουν την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται ώστε ο καθένας να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του και να αποφύγουμε καταστάσεις παράλογες όπου έχουμε ισχυρή ε, γεωργική βιομηχανία αλλά δεν είναι καλά αμοιβόμενο ούτε ο γεωργός ούτε ο καταναλωτής ο οποίος πληρώνει ένα προϊόν το οποίο να είναι ισορροπημένο αν θέλετε σε σχέση με αυτά τα οποία πληρώνει για να αποκτήσει. Γι' αυτό η οργάνωση των παραγωγών, η μελέτη της αγοράς και η συνδυασμός διαφόρων στοιχείων θα είναι απαραίτητα για να κάνουμε καινοτομίες όχι μόνο για την παραγωγή αλλά και για την οργάνωση που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ των φιλοδοξιών για παραγωγή και είδαμε εδώ ότι το θέμα της παραγωγικότητας τίθεται και πρέπει να βρεθούν μέσα ώστε η αύξηση της παραγωγικότητας να μην γίνει εις βάρος της βιωσιμότητας της γεωργίας και βεβαίως τα μέτρα που προτείνονται στην μεταρρύθμιση δεν είναι επαρκή, δεν είναι τέλεια ίσως, αλλά πρέπει να έχουν την φιλοδοξία να δημιουργήσουν κίνητρο ώστε να πάρει κάποια άλλη κατεύθυνση η γεωργία μας. Επίσης, υπάρχει η προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων ανατόπο. Θέλω να επαναλάβω ότι εμεί δεν προτιθέμεθα από τις Βρυξέλλες να αποφασίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό στη θέση των κρατών μελών τι κάνουμε. Δημιουργούμε ευκαιρίες και δυνατότητες τις οποίες μετά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εποφελώς οι... τα κράτη, οι κυβερνώντες, οι υπεύθυνοι πολιτικές, οι επαγγελματικές οργανώσεις. Μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε και να εξαγγείλουμε όποιο μέτρο θέλουμε. Αλλά εάν δεν είναι σαφές ότι αυτά που λέμε θα γίνουν με προσαρμογή στα εθνικά μέτρα, δεν θα έχουμε μια ισχυρή πολιτική ανάπτυξη τη υπαίθρου. Τελειώνοντας, θα πω το εξής. Αυτή η γεωργική πολιτική δεν είναι επαρκής, αλλά είναι απαραίτητη για να δώσουμε ένα νέο προσανατολισμό στις φιλοδοξίες του κλάδου για την ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους σήμερα μας προσέφεραν τις αναλύσεις τους, τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους. Αυτό είναι σημαντικό στα πλαίσια της διαδικασίας που ακολουθούμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κάθε φορά μας υποδέχεται με ανοιχτό πνεύμα και αναμένοντας πολλά από αυτές τις συναντήσεις και θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία με εσωτερικέ συζητήσει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στη διαδικασία, αλλά και τη διάρκεια όλου του έτου 2012 θα συνεχίσουμε να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ώστε κάθε φορά να έχουμε το feedback πριν να λαμβάνουμε τι αποφάσει. Ανοιχτά λοιπόν είναι τα πάντα προ την κοινή γνώμη. Και τελειώντα θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά και του διερμηνεί που κάθε φορά μας αντιμετωπίζουν με μεγάλη ενεργητικότητα και υπομονή ώστε να μπορέσουμε ο καθένας στη γλώσσα του να πει αυτό που πρέπει να πει ώστε στο τέλος όλοι να καταλάβουν.